Colleagues, good afternoon Καλησπέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους και την πρόεδρο Σατόρη από την Επιτροπή Ήτρε και τα μέλη της Ήτρε στην Επιτροπή Μεταφορών για τη συνεδρίασή μας την απογευματινή είναι μια κοινή συνεδρίαση. Αφορά το χρηματοδοτική διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Πριν σας δώσω το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, σας ε, Προέδρε και τη Γραμματεία για τη στενή ε, συνεργασία μας. Απολαύσαμε αυτή τη συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό η Ήτρε και η Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών να συνεργαστούν σε αυτό το θέμα και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία με εσάς και τους συναδέλφους σας. Υπάρχει ξεχωριστή ημερήσια διάταξη για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, συνάδελφοι. Οπότε αυτήν να ακολουθώ να σας υπενθυμίσω ότι εδώ ακολουθούμε το άρθρο 51 του εσωτερικού κανονισμού. Βάσει αυτού κινούμεθα. Με βάση αυτό το άρθρο ε, κινούμαστε και συνεργαζόμαστε και οι συγγητές μας και οι συγγητές σας συνεργάζονται και αποστέλουν μία έκθεση ε, στο Κοινοβούλιο προς εξέταση. Συνήθως συμπροεδρεύουν οι δύο πρόεδροι των Επιτροπών σε αυτές τις συνεδριάσεις, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ και οι δύο, για να διευκολύνουμε τη διαδικασία, συμφωνήσαμε ότι ο πρόεδρος της, ε, της, του οικοδεσπότη της Επιτροπής που φιλοξενεί είναι πρόεδρος, ο πρόεδρος. Ε, έχουμε εμείς την Τραν που προεδρεύει. Όταν πάμε στην, έχουμε τη μεικτή συνεδρίαση και μας φιλοξενεί η Ήτρε θα προεδρεύει η κυρία Σαρτόρη. Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να ε, πάρει το λόγο. Παρακαλώ να δείξετε ενδιαφέρον να μιλήσετε και θα σας αφήσουμε να παρέμβετε. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Σατόρη να κάνει κάποια αρχικά σχόλια και μετά από αυτό θα απευθυνθώ προς συνεισηγητές. Λοιπόν κυρία Πρόεδρε Σατόρη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε όλοι. Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Ήτρε ακολουθεί αυτή τη διαδικασία του άρθρου 51 και γι' αυτό για μας ως Επιτροπή αυτή είναι μια εμπειρία. Η σημασία της προτάσεως που αφορά τους μηχανισμούς για τη σύνδεση της Ευρώπης ε, είναι κάτι που δικαιολογεί αυτή την κοινή συνεδρίαση και χάρη στα αποτελέσματα των εργασιών μας πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις που θα βοηθήσουν να υλοποιήσουν στρατηγικούς στόχους στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών, της ενεργείας και του, των μεταφορών. Όλα αυτά ε, δικαιώνουμε την εκείνη συνεδρίαση. Τις τελευταίους μήνες συνεργαστήκαμε οι πρόεδροι και ελπίζω ότι και μετά από αυτή την ημέρα θα συνεχιστεί η συνεργασία μας και μάλιστα θα βελτιωθεί. Και εύχομαι καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Σατόρη είμαι σίγουρος ότι αυτό πράγματι θα γίνει, πρώτα θα καλέσω τον Γκόραν Φάρμ της Επιτροπής Προϋπολογισμών να πάρει το λόγο, διότι όλοι υπακούμε την Επιτροπή Προϋπολογισμών και τη σεβόμαστε, ε, εσύ και μετά θα ακούσουμε τους εισηγητές, την κυρία Βαριένα από την Ήτρε, ο κύριος Ρικέ και η κυρία Γιάλα Σάντερ θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, Γκόραν, θα ξεκινήσουμε με εσένα για να μπορέσει να μας κρατήσει έτσι μαζεμένους θα είμαι σχετικά σύντομο, λέει ο Γκόραν. Δεν έχω πολλά να πω όσον αφορά το θέμα αυτό καθε αυτό, διότι ακόμα και αν είμαι εισηγητή για την Επιτροπή Προπολογισμών για τι υποδομέ, ξεκινήσαμε τι συζητήσει βασικά πάνω σε ένα κομμάτι αυτό που είναι τα οικονομικά μέσα, κυρίω όσον αφορά τα ομόλογα έργων και έχουμε εκπονήσει μια έκθεση για την πρωτική φάση αυτών των ομολόγων έργων αλλά βεβαίω θα διεξαχθεί και ευρύτερη συζήτηση για τη χρήση των χρηματοστικών μέσων όσον αφορά το μέσο για την ε, σύνδεση τη Ευρώπη που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τώρα συντονίζουμε τι διαπραγματεύσει του προπολογισμού ή μάλλον τι διαπραγματεύσει του δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι δημιουργήσαμε ε, μια ομάδα επαφή στο Κοινοβούλιο υπό την ηγεσία του Μάρτιν Σούλτ, του Προέδρου, και με τη διαπραγματευτική ομάδα για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τους συντονιστές τη Επιτροπής Προπολογισμών κινούμεθα, αλλά και σε αυτή την ομάδα επαφών όταν χρειάζεται θα συμπεριλαμβάνουμε και ε, εκπροσώπους των καθήλων αρμοδίων επιτροπών και έγινε σήμερα συνεδρία της ομάδας ε, επαφής οπότε συζητούμε πώς μπορούμε να συντονίσουμε τους ρόλους των ειδικών επιτροπών σε πάνω από τα 60 νομικά μέσα τα οποία διαπραγματευόμαστε και στο Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα συντονίσουμε σε διαπραγματευτική θέση για το οικονομικό πλαίσιο στο σύνολό του. Εγώ, α, μάλλον η ομάδα επαφής πρότεινε να επεξεργαστούμε στο βαθμό του δυνατού στο Κοινοβούλιο και σε επίπεδο επιτροπών το θέμα να προχωρήσουμε όσο γίνεται χωρίς να πάμε στην Ολομέλεια να αποφασίσουμε επί στοιχείων αριθμητικών μέχρι ότου γνωρίζουμε τι του Συμβουλίου και γνωρίζουμε τότε το Συμβούλιο θα παρουσιάσει, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα κουτί πακέτο διαπραγματεύσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος Ιουνίου όπου εκεί θα παρουσιαστούν διάφορες κοινέ θέσεις των κρατών μελών και του Συμβουλίου επί όλων των θεμάτων. Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα προχωρήσουν, σε πόσες λεπτομέρειες θα μπουν, αν θα αναφέρουν στοιχεία αριθμητικά ή μόνο τις αρχές και μετά θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μετά το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι αν όλα πάνε καλά, αλλά σε υπενθυμίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο. Διότι διάφορα κράτη-μέλη και σημαντικά κράτη-μέλη αποφάσισαν ότι η πολιτική τους είναι η περικοπή κατά 100 δις ευρώ για την επόμενη θετία του όλου πλαισίου, περικοπή δηλαδή του 10% του δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό βεβαίως αν παραμείνει η θέση του Συμβουλίου θα δημιουργήσει τεράστιες δυσκολίες για μας για να επεκτείνουμε οι εσδήποτε πολιτικές όσο και καλά επιχειρήματα να έχουμε αυτές τις πολιτικές. Αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες που σας δίνω όσον αφορά τις και βέβαια είναι σημαντικότατο σε αυτή την κατάσταση να συμφωνήσουμε επί των βασικών προτεραιοτήτων. Και αυτό που τονίζουμε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις είναι ότι χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό για επενδύσεις. Επενδύσεις για ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα που έχουμε. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα για να υπερασπιστούμε τον προϋπολογισμό στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Και βεβαίως και το μέσο αυτό για τη σύνδεση της Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσο για τις επενδύσεις και χρειάζεται χρηματοδότηση. Αυτά ήθελα να πω εν είδη εισαγωγή. Ε, διαφορετικά πρέπει να σας πω ότι είμαι εδώ για να ακούσω τι θα πείτε. Σας ευχαριστούμε κύριε Φάρμ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Βαλιάν, που είναι η συγκήτρια της Επιτροπής Βιομηχανίας της ΙΤΡΕ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο ε, η συγγήτρια της Ήτρε για τη διευκόλυνση αυτή ε, συνδέοντας στην Ευρώπη σε αυτή την πρώτη κοινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια της Επιτροπής Μεταφορών, Αγιάλα Σέντερ και Ντομινίκ Ρικέ, ε, για τις πολύ χρήσιμες συναντήσεις και καρποφόρες ε, συνομιλίες που είχαμε. Έχουμε τρεις εισηγητές για το ίδιο θέμα, από οργανωτική άποψη μεγάλη πρόκληση. Η διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη είναι ένα νέο θέμα, ένα νέο κοινοτικό ενωσιακό μέσο και καλό θα ήταν να, κάνουμε μια σύντομη παρουσίασή του στους συναδέλφους ε, για τον προφανή λόγο να τους ε, ε, ενημερώσουμε και το θέμα αυτό. Είναι ένα σχέδιο με 500 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις για τη βελτίωση των ενεργειακών ε, ε, μεταφορικών και ψηφιακών δικτύων. 31,7 δισεκατομμύρια θα χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση των υποδομών ε, δημιουργία, ε, γεφύρωση των κενών και αποσυμφόρηση. 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής για σχέδια μεταφορών στις χώρες συνοχής και 21,7 δισεκατομμύρια θα διατεθούν στα κράτη-μέλη για τις επενδύσεις ε, σε μεταφορές, σε υποδομές μεταφορών. 9,1 δισεκατομμύρια θα αφιερωθούν στον ενεργειακό τομέα για τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του 2020 για την ενέργεια, ε, τις κλιματικές αλλαγές. 1,2 ε, θα έχουμε δισεκατομμύρια επενδύσεις για ψηφιακές υπηρεσίες και τα ομόλογα έργου που προτείνονται είναι ένα τμήμα του συνολικού πακέτου του συνδέοντα στην Ευρώπη, προκειμένου να δημιουργηθεί μια μόχλευση των ιδιωτικών και κρατικών κονδυλίων για να δοθεί προβολή σε ορισμένα προγράμματα και να μειωθεί ο κίνδυνός τους. Η νέα διευκόλυνση αυτή, το συνδέοντα στην Ευρώπη, θα πρέπει να ε, θεωρηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου του 2014-2020 και των σχετικών διαπραγματεύσεων. Αυτό το νέο χρηματοδοτικό αρχιτεκτόνιμο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στόχο έχει να υλοποιήσει τη στρατηγική του 2020 και τροποποιεί την προσέγγιση προσπαθώντας όχι μόνο να εξασφαλίσει ε, υγιή προϋπολογισμό αλλά να υλοποιήσει τους στόχους χάρη στη συνέργεια και την ε, ανταγωνιστική ανάπτυξη. Η συνέργεια βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ουσιαστικά αποτελεί την πεπτουσία τη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη Αξία. Θα πρέπει όπου μπορούμε να πλουστεύουμε τα προγράμματα και να προβαίνουμε σε ενοποίηση των τομεακών πολιτικών. Αυτό το μέσο ιδέοντα την Ευρώπη συνιστά την πρώτη καλή απόπειρα προ την κατεύθυνση αυτή. Βέβαια, οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε είναι και χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα. Οι χρηματοπιστωτικέ αδυναμίε, τα ελλείμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν διορθωθεί από τα επιμέρου μέτρα που λάβαμε μέχρι στιγμή ε, και δεν ε, αντιμετωπίζουν τα αίτια των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Χρειάζεται φυσικά δημοσιονομική ε, ισορροπία και πειθαρχία για να μπορέσουμε να εφαρμόζουμε τις βιώσιμες πολιτικές μας. Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε σήμερα ένα πρόσφορο για την αντιγωνιστικότητα κλίμα και για την ευφυή ανάπτυξη, προκειμένου να διορθώσουμε ένα σύστημα που αποδείχθηκε ότι δεν είναι βιώσιμο. Και παρά τον την πρωτογενή ανάπτυξη βασικών τομέων της οικονομίας. Οι υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φαίνεται ότι γίνονται όλο και πιο απερχιωμένες και δεν υπάρχει επαρκής διασύνδεση μεταξύ τους. Ο κατακαιρματισμός της αγοράς και η επανεθνικοποίηση των πολιτικών στον τομέα της ενέργειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών είναι σημαντικές απειλές ε, της ε, σημερινής είναι σημαντικές απειλές αν το, η, η μέχρι τώρα προσέγγιση διονυστεί. Ε, δεν έχει νόημα να πούμε στο φαύλο κύκλο να περιμένουμε επενδύσει που δεν έρχονται ποτέ. Είναι η ευκαιρία να φανούμε καινοτόμοι και ευρηματικοί στη, στο νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Βέβαια, θα χρειαστούν κάποιε προσπάθειε για να υλοποιήσουμε του στόχου τη στρατηγική του 2020 για τα ενεργειακά δίκτυα 500, για τι μεταφορέ, 200, για, για τις τηλεπικοινωνίες και, και την πληροφορική δεν μπορούμε λοιπόν να επιδοψηλεύουμε κονδύλια κρατικά σε μαζικά προγράμματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ιδιωτικές επενδύσεις και να κάνουμε τη, τα κοινωτικά προγράμματα ελκυστικά και για τους ιδιώτες για να επενδύσουν. Επίσης χρειαζόμαστε μια βιωσιμότητα και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η διευκόλυνση δέντος της Ευρώπης θα πρέπει να στηρίζεται σε διαφανείς διαδικασίες και προτεραιότητες που θα εξασφαλίσουν ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, κάτι που είναι απαραίτητο για τους ιδιώτες επενδυτές ε, κάποιοι θεσμικοί επενδυτέ, όπως στα εξωτερικά ταμεία και οι ασφαλιστικέ εταιρείες έχουν μέσα και κονδύλια να επενδύσουν αρκεί να σταματήσει ο θέμητο ανταγωνισμός μεταξύ της κρατική και της ιδιωτικής επένδυσης. Ε, το μέσο αυτό ιδιαίτερα στην Ευρώπη μου είπαν ότι ε, θα περιλαμβάνει τα κονδύλια που θα αφιερώσει στις υποδομές Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ διαφωνώ γιατί η ιδέα του κοινού εργαλείου του κοινού μέσου για την χρηματοδότηση των υποδομών στην Ευρώπη προϋποθέτει μια, ένα συντονισμό των προτεραιοτήτων των πολιτικών και μια σωστή εφαρμογή. Το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη είναι πρώτα απ' όλα ένα εργαλείο που θα φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά σε μια εύρυθμη λειτουργούσα εσωτερική αγορά που θα ε, προωθεί την ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργεί τη βάση για την ανάπτυξη. Στη φάση αυτή ευελπιστώ ότι θα το πετύχουμε, αλλά θα είμαι και κριτική ταυτόχρονα. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τον εαυτό όργανο, δεν θα πρέπει να το δεχτούμε ε, ανεφόρον. Επίσης, δεν θα πρέπει να επηρεάσουμε αρνητικά την αγορά με κάποιες παρεμβάσεις μας, ούτε θα πρέπει να αποτρέπουμε ε, τους επενδυτές ή να δημιουργούμε στρεβλώσεις. Οποιοδήποτε δαπάνη θα πρέπει να εξετάζεται υπό το φως σαφών κριτηρίων, που θα λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις ανησυχίες. Είναι πραγματικά καινοτόμο ο χαρακτήρα αυτού του νέου χρηματοδοτικού οργάνου. Γι' αυτό και ε, καταλαβαίνω την επιφυλακτικότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το προκαθορίσει πώ θα ξοδεύονται τα κονδύλια και θα πάνε. Αλλά οι αγορέ γενικώ ε, αντιδρούν αρνητικά σε κάποιε αόριστε και απροσδιορίστε δηλώσει. Πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να έχουμε διαβούλευση με φορείς της πραγματικής οικονομίας και αγοράς, ώστε να επικεντρώσουμε αυτό το μέσο στις συγκεκριμένες ανάγκες των αγορών τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και ενέργειας. Και ο λόγος μεταξύ επιχορηγήσεων και ιδιωτικής και κρατικής χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να αφαιθεί για εκ των υστέρων διευθέτηση, γιατί θα δημιουργήσει πάλι έναν ε, επενδυτικό μηχανισμό που δεν θα ελκύει τους επενδυτές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να διαιρούμε τεχνητά κάποια επενδυτικά μέσα που δεν θα ελκύσουν τους επενδυτές. Χρειαζόμαστε καλή επικοινωνία, συνδρομή, απλούστευση και αξιοπιστία. Αυτό δείχνει τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το περίπλοκο θέμα που για, για το οποίο χρειάζονται πολιτικές αλλά και τεχνικές δεξιότητες. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τους δύο συνεισηγητές, Σέντερ και Ρικέ, με τους σκιώδες συνεισηγητές επίσης και με όλους τους ε, συναδέλφους ε, που ενδιαφέρονται από τις Επιτροπές Ρέτζι, Προπολογισμών, ε, Ήτρε, Τραν και τώρα θα δώσετε φαντάζομαι το λόγο στους συνεισηγητές της Επιτροπής Μεταφορά και Τουρισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βαλιάν. Τώρα θα ακολουθήσουν οι δύο εισηγητές των μεταφορών. Πρώτα ο κ. Ρικέ. Θέλω να... και μετά κύριε Σέντερ. Θέλω να ακούσω βέβαια και τους άλλους. Μάικλ, ναι, εσύ πάντα θέλεις να μιλήσεις. Σε έχω γράψει λοιπόν ήδη. Πρώτο ο αντιπρόεδρος μας κύριος Ρικέ και μετά θα ακολουθήσει η Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ήτρε. Σημαντική για μένα ικανοποίηση να συνεργαστώ με δύο κυρίες εισηγήτριες. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά και βέβαια το θέμα είναι περίπλοκο ε, και ο τρόπος συνεργασίας είναι περίπλοκος. Πρώτα εκφράζω την ικανοποίησή μου για την τολμηρή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θέτει ορισμένα προβλήματα και να πω ότι για την ώρα ως έχει το θέμα υπάρχουν αυτές οι τρεις οδοί προσέγγισης που προσφέρει αυτό το μέσον και τα τέσσερα προβλήματα που θέτουν και που είναι η ουσία της κοινοβουλευτικής εργασίας. Η τριπλή προσέγγιση της CEF είναι η συγκέντρωση, η απλούστευση και η τεχνική υποστήριξη. Η συγκέντρωση δεν είναι βέβαια μόνο των δικτύων, είναι και η οργάνωση σύμφωνα με τη διάκριση σε κεντρικά και περιφερειακά δίκτυα, η διάδρομη, το πέρασμα από πετρέλαιο σε δίκτυο και θέματα ορατότητας και λειτουργικότητας που πρέπει να βελτιωθεί. Δεύτερο, πρόκειται για απλοποίηση ευθυγράμμιση δηλαδή των δικτών της στρατηγικής 2020 με το παρόν μέσον που θα δώσει μια ευκαμψία στα κονδύλια, στα κοινά μέσα και στις κοινέ χρηματοδοτήσεις. Το κείμενο βασίζεται στις συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν ανάμεσα στον τομέα των μεταφορών της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών βασισμένο στην ιδέα ότι οι προβληματισμοί είναι παρόμοιοι και ότι μια κοινή διαχείριση θα ήταν καλύτερα για όλους και για την εφαρμογή αλλά και για την συνέχεια. Και τέλος το τρίτο είναι το εργαλείο της τεχνικής υποστήριξης γιατί στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια πραγματική εμπειρογνωμοσύνη και αυτή η τεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη για το ΣΥΕΦ e γιατί είναι δύσκολα και περίπλοκα τα χρηματοδοτικά μέσα Μιλούμε πάντα για την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, για την χρήση κονδυλίων που προέρχονται από διάφορες προελεύσεις και ορισμένες φορές και από το Ταμείο Σύνοχης και το τεχνικό μέρος επί της ουσίας, αλλά και για το χρηματοδοτικό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης, συγκεντρωτικής προσπάθειας αν θέλετε. Καλύτερη λοιπόν αποδοτικότητα, καλύτερη αποτελεσματικότητα διότι συγκεντρώνονται οι προσπάθειες, απλουστεύονται όλοι οι φάκελοι αυτοί και δημιουργούνται συνέργειες. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα. Έχω εντοπίσει τέσσερα που αντιστοιχούν και στα μεγάλα κεφάλαια των δυσχεριών αυτών. Πρώτα-πρώτα η χρηματοδοτική πτυχή. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει σχετικά σύντομα για τις λεγόμενες guidelines, όταν όμως φτάσουμε στη χρηματοδότηση, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ και για το Κοινοβούλιο αλλά και ιδίως για το Συμβούλιο. Όπως είπε σωστά ο Γιώραν Φέρμ, η διευκόλυνση συνδέτα στην Ευρώπη είναι ένα από τα κουτιά μέσα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και είναι δύσκολο να απομονωθεί ε, το κουτί αυτό. Αυτό βέβαια θέτει και το θέμα των ποσών που ανέφερε ο Γιώραν Φέρμ οι, τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών λένε όχι, προσοχή, όχι ακόμα, μην γράψουμε ακόμα νούμερα γιατί μπορεί να διαλυθεί όλο το πλαίσιο αυτό. Βέβαια το, η ουσία είναι ξεχωριστή από τα κονδύλια. Αν όμως είναι για παράδειγμα 50 δισεκατομμύρια, διαφορετικό από όταν το ποσό πολύ χαμηλότερο και υπάρχουν και άλλα προβλήματα δημοσιονομικά εκτός από το απόλυτο νούμερο που είναι δηλαδή οι διαφορετικές προελεύσεις των κονδυλίων ιδιαίτερα από το Ταμείο Συνοχής με την ιδιαίτερη αυτή περιφερειακή διαχείριση ε, της οποίας χαίρει και βέβαια κυρίως που είναι για τις ε, χώρες της συνοχής. Το άλλο πρόβλημα είναι της διάθεσης των κονδυλίων, του προορισμού των κονδυλίων. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα από όλες τις πλευρές, διότι με ένα μηχανισμό σαν αυτό έχουμε κατανείμει τα κονδύλια ανάμεσα στα έργα, ανάμεσα στους μηχανισμούς χρηματοδότησης και ανάμεσα στις πηγές χρηματοδότησης. Το σύνολο αυτών των τριών αξώνων πρέπει τελικά να ε, λειτουργήσει. Μέσα από τα διάφορα σχέδια και τον καθορισμό των διαδρόμων πρέπει να γίνει και η διάκριση ανάμεσα σε παλαιά έργα, νέα έργα κλπ και ο μηχανισμός των χρηματοδοτήσεων θα πρέπει να είναι ξεχωριστά για τις επιδοτήσεις γνωστά μέσα χρηματοδότησης, καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης. Βέβαια μπαίνουν στη μέση και οι εγγυήσει, τα ομόλογα έργων και η μεικτή χρηματοδότηση. Επομένως δεύτερο επίπεδο διάκρισης και τρίτο επίπεδο διάκρισης ανάμεσα στις πηγές χρηματοδοτήσεων των διαφόρων ταμείων, ταμείων συνοχής κλπ. Τι μπορεί να προσφέρει το ένα ταμείο, τι μπορούν να προσφέρουν άλλοι οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τι μπορούν να προσφέρουν οι ιδιωτικοί φορείς. Και πρέπει λοιπόν να αποκατασταθεί και τελικά μια ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο χρήμα και στο ιδιωτικό χρήμα. Δηλαδή πρόκειται για την δημοσιονομική διαχείριση των έργων, άρα πρέπει να επιλεγεί το έργο, ο μηχανισμός της χρηματοδότησης και βέβαια και η προέλευση των κονδυλίων. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να ενταχθούν μέσα στο συνολικό μηχανισμό. Και το τρίτο είναι η διακυβέρνηση, η governance, που είναι βέβαια ευρωπαϊκή, κοινοτική, αλλά με ποια κατανομή μεταξύ κομισιών, εκτελεστικών οργανισμών, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που είναι και αυτό από τα θεσμικά οργανά της Ένωσης, ποιος είναι ο ρόλος της επιτροπολογίας και βέβαια εν τέλει και πώς εμπλέκονται το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών, πώς ενημερώνονται και πώς διατηρούν την αρμοδιότητα ελέγχου. Και στο εθνικό επίπεδο πρέπει να αναρωτηθεί κανείς ποιον ρόλο θα αναλάβουν οι χώρες μέλη και κυρίως για τα κονδύλια που έρχονται από τα Ταμείο Συνοχής, πώς θα διαθέσουν τα δικά τους κονδύλια, ποια είναι η δυνατότητα να συζητηθούν τα έργα αυτά σε περιφερειακό επίπεδο και τέλος οι διάδρομοι που είναι επίσης ένα αντικείμενο συζήτησης και πρέπει να μην θεωρηθούν απλά σαν κατευθυντήριες γραμμές, σαν γεωγραφική επιλογή αλλά και σαν εργαλείο διακυβέρνησης. Ε, περαιώνω εδώ για να πω ακόμη ότι η πρόκληση θα είναι βέβαια να λάβουμε τελικά και τα κονδύλια από το Συμβούλιο. Να καταφέρουμε να κατευθύνουμε σωστά τις προσπάθειες όλων των διαφόρων ε, μερών, χωρών μελών, ε, θεσμικών οργάνων κλπ. Να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της Ένωσης και βέβαια είναι το ωραιότερο έργο ανάπτυξης αυτό για την Ευρώπη, για την απασχόληση, για τον ανταγωνισμό, για την ανταγωνιστικότητα μάλλον και πραγματικά είναι μια τεράστια πρόκληση αλλά αξίζει να αγωνιστεί κανείς για αυτήν. Ευχαριστώ κύριε Γιάλα Σέντερ τώρα και έχω ένα μακροσκελή κατάλογο αγόριτων και δεν έχουμε και τελείω το χρόνο να το έχετε υπόψη. Κύριε Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ φυσικά να καλωσορίσω την κυρία Σαρτόρη, την κυρία Βαλεάν και όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας, τη ΣΥΤΡΕ. Νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία της συνεργασίας μας γιατί στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε ένα νομοθετικό κείμενο που θα βοηθά μεταξύ άλλων ε, την πρόθεση της συνέργειας μεταξύ τριών βασικών αξώνων. Φυσικά τώρα βρισκόμαστε στο γενικό πλαίσιο, στο πρώτο στοιχείο και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και το χρονοδιάγραμμα και στην παρούσα ε, κρίση, τη χρηματοπιστωτική και την οικονομική στην Ευρώπη και με τις απαιτήσει των Ευρωπαίων πολιτών να αντιμετωπιστούν ε, η ανάπτυξη, να γίνουμε ανταγωνιστικοί προς την Κίνα και τους άλλους εταίρους. Η ανταγωνιστικότητα είναι θέμα σημαντικό. Οπότε ε, η ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά της ε, διευκόλυνσης αυτής του συνδέοντας στην Ευρώπη. Και φυσικά καλύτερη προβολή όλων των προσπαθειών υπέρ της ανάπτυξης. Όπως είπε ο κύριος Φάρμ, έχουμε το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και πλησιάσει ο καιρός των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Ε, και φυσικά έχουμε τις ε, τα αιτήματα όχι μόνο των συναδέλφων της Επιτροπής Προϋπολογισμών αλλά και του Συμβουλίου γενικώ, αλλά και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής μερικές φορές το αίτημα να μην ε, ε, αναφέρουμε στοιχεία αριθμητικά αλλά μόνο αρχές. Με την διευκόλυνση όμως του συνδέοντος στην Ευρώπη το μόνο στοιχείο που έχουμε είναι ότι ουδέποτε δεν είχαμε επαρκή χρηματοδότηση για να μπορέσουμε πραγματικά να επικεντρωθούμε στην αποσυμφόρηση, στις στενοπούς εκείνες ε, να τους, να τους εξελίψουμε ώστε να έχουμε πραγματικά προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο, να τονίσουμε την ελληπή χρηματοδότηση, χωρίς να φέρουμε συγκεκριμένα νούμερα, αλλά να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα κονδύλια για να ξεφύγουμε από το μαρασμό που μας βήθησε η προηγούμενη ε, απόφαση για τις δημοσιονομικές προοπτικές, για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη ε, και τις επενδύσεις υποδομές, ψηφιακές, ενεργειακές ε, και μεταφορές και να μην περικόψουμε κονδύλια εκεί. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συνέργεια, εκεί είναι που έχουμε πολύ μεγαλύτερο περιθώριο να αναπτύξουμε τις διασυνδέσεις μεταξύ των τριών αξώνων ανάπτυξης που είναι οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και η ενέργεια. Και φυσικά ανέκαθεν λαμβάναμε υπόψη αυτές τους τρεις άξονες γιατί στην Επιτροπή Μεταφορών ασχολούμασταν και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις νέες απαιτήσει για τους νέους τρόπους ενέργειας και φυσικά θα πρέπει με ευφύ τρόπο να βελτιώσουμε τα συστήματα μεταφορών. Τώρα, για την διευκόλυνση αυτή του συνδέοντος στην Ευρώπη, την ΕΦΣΥ, στόχος μας ε, είναι να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Βέβαια, το Συμβούλιο μας έκανε ένα δώρο άδωρο ουσιαστικά, γιατί στις πτυχές που θέλαμε να επιμείνουμε εμείς, που ήταν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, εκείνη ακριβώς που το Συμβούλιο ε, χαρακτηριζόμενο από μία σπουδή και βιασύνη που δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε το λόγο της και με τις περίεργες αυτές τρόικες και τις συμφωνίες τους καταλήξαμε ε, σε ένα περισσότερο διακυβερνητικό μέσο παρά σε οτιδήποτε άλλο πανευρωπαϊκό δηλαδή όπως επιθυμούσαμε εμείς. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να ενισχύσουμε την πανευρωπαϊκή διάσταση, την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτός είναι βασικός ε, στόχος μας. Και φυσικά να εξασφαλίσουμε συνέργεια μεταξύ του Ταμείου Συνοχής και των Ταμείων των Διευρωπαϊκών Δικτύων. Αυτό να φαίνεται στην κατανομή ε, των κονδυλίων μεταξύ των ε, κρατών συνοχής και των υπόλοιπων και φυσικά να επικεντρωθούμε στην σωστή εφαρμογή και αξιοποίηση των κονδυλίων. Επικεντρωνόμαστε επίσης σε διαδρόμους. Είναι όργανο διακυβέρνησης αλλά και όργανο ε, διαχείρισης και έχουμε φυσικά τα βασικά δίκτυα αλλά μας ενδιαφέρουν και τα διάφορα εργαλεία της χρηματοδότησης και θα έχουμε και το νέο ρόλο του εκτελεστικού οργανισμού που θα mm. μας εξασφαλίσει την εκτέλεση στα πλαίσια των τριών αξώνων που αναφέραμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιαλασέντα. Θα δώσω το λόγο σε εκείνους που θέλουν να μιλήσουν, να μαζέψω στον κατάλογο και θα μοιράσω το χρόνο ισότιμα. Got Mr. Kanchan, Mr. Perillo, Mr. Tobacco, Mr. Kramer, Zeal, Mr. Vidal, Mr. Alcadrawe, Mr. Gross, Mr. Koumoutsakos, Mr. Bradbourne. Mrs. Tikal,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 θα ήθελα να ξαναδιαβάσω τον κατάλογο, με αυτούς θέλω να πάρουν το λόγο. Θα τον κλείσω τον κατάλογο, αλλιώς όλοι τελικά θα έχουμε μόνο 30 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι τα ονόματα εκείνο που έχουν ζητήσει στο λόγο. Είστε όλοι ικανοποιημένοι. Ακόμα ανοιχτό ο κατάλογο. Τέρμα. Κατακυρώθηκε, έκλεισε. 14 θέλω να πάρω το λόγο. Επί τρία λεπτά ο καθένας. Ένα τρίλεπτο, παρακαλώ. Ξέρουν ότι απειλώ με σφυριά ε, τα μέλη της Επιτροπής ε, Μεταφορών. Ο κ. Καντσάν έχει πρώτος το λόγο και είναι ο πρώτος που θα απειληθεί με σφυριά αν πάει να ξεπεράσει το χρόνο που του διατίθεται. Πρέπει να είστε πιο ανεκτικός με μένα, διότι είμαι σκιώδης ηγητής για το θέμα αυτό του μέσου τη συνδέοντα την Ευρώπη και σαν μέλος Επιτροπής των Μεταφορών έχω κάτι να πω έτσι. Ε, η... Το μέσο αυτό συνδέοντα την Ευρώπη, η επένδυση, ανάπτυξη, απασχόληση, όλα αυτά είναι μια σειρά διασυνδέσεων και διαθρώσεων που στην πραγματικότητα όμως δεν βλέπω πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Συνοψίζω την παρέμβασή μου σε τέσσερα σημεία να διατηρηθεί το κονδύλι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άκουσα τον πρώτο εισηγητή που ήδη είπε ότι ένα μείον 10% είναι ήδη επιτάπητος. Δεύτερον, εξορθολογισμός εκείνο που έχουμε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το μείγμα των δύο επιτροπών, Ρέτζι και Τραν, για να προσπαθήσουμε μαζί να ε, μαζέψουμε τα 10 δισεκατομμύρια και μας φεύγουν από τα δάχτυλα τα λεφτά. Θα πρέπει ε, να δώσουμε κάποια κίνητρα και να φροντίσουμε εκείνος που κάνει τον προγραμματισμό των δικτύων και να έχει κίνητρα. Εξορθολογισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάω προς το, στο σημείο, προς τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης. Είχαμε σήμερα τα project bond το πρωί, τα συζητήσαμε, είναι ένα μέσο που θεωρούμε ότι είναι μικρή θεραπεία, σαν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε μέσα σπυρίνη στον ασθενή. Ε, διαθέτουμε πολύ μικρά κονδύλια για να εγγυηθούμε επενδύσεις ε, που κάνουν οι εταιρείε των έργων. Τέταρτο, είναι κάτι που πιστεύω και θέλω να ακούσω απαντήσεις από τους συναδέλφους διότι ήρθε η στιγμή να το συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα, να ακούσουμε ναι ή όχι, να ξεπεράσουμε τα του προπολογισμού. Ένα το σύστημα ε, εταιρικών σχέσεων με και διαφόρων συν, ε, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να έχουμε το θάρρος να προχωρήσουμε πιο πέρα από το μέσο αυτό που θέλουμε να διαθέσουμε στη σύνδεση της Ευρώπης και τα συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πρέπει να προχωρήσουμε πιο πέρα. Να διαθέσουμε ομόλογα, δεν ξέρω, μπόντα τα πούμε σκέτα, για να συνεννοούμεθα, δεν ξέρω πώς θα τα αποκαλέσουμε. Και αυτά τα χρήματα και αυτά τα ομόλογα άμεσα να μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση των υποδομών, των έργων υποδομών, από μεταφορέ, για ενέργεια, για τηλεπικοινωνίες, όλα αυτά. Ε, 1.500 εκατομμύρια έχουν διαθέσει. Συμφωνούμε ότι είναι καλή στιγμή ε, για να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ή μένουμε δεσμευμένοι όσον αφορά αυτό το μέσο για τη σύνδεση της Ευρώπης και στα πλαίσια του προπολογισμού. Αυτό είναι το ερώτημα που έχω και θα ήθελα κάποιος να δώσει μια απάντηση. Ή να πει ότι δεν έχω σχόλιο ή να πει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Αλλά κάναμε τόσα πολλά. Ξεπεράσουν τι συνθήκε όσον αφορά τη λιτότητα. Νομίζω ότι και αυτή η, μορφή που, αυτή η φωνή που συνδέεται με την ανάπτυξη είναι κάτι που συνδέεται με αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ε, με αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας στον περιπολογισμό να πετύχουμε την ε, ανάπτυξη. Σας έδωσα λίγο παραπάνω κύριε Κάντσα, λέει ο Πρόεδρος. Ο Πυρίλο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε ένα πακέτο για τις υποδομές, για τις μεταφορές, την ενέργεια, για τις τηλεπικοινωνίες. Σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα είναι βασικό παράδειγμα για την επίτευξη πραγματικής εσωτερικής αγοράς. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, χρειάζεται να ξανασκεφτούμε την ευρωπαϊκή στρατηγική στα πλαίσια των υποδομών. Για πολλά χρόνια αυτό αφέθηκε στα κράτη-μέλη να το κάνουν, αυτόνομη στρατηγική επενδυτική, που ποτέ δεν είχε συντονιστεί από ένα ρυθμιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό ευνόησε την προστασία των συμφερόντων κάποιων κρατών μελών με κάποια ωφέλη σύντομα. Αλλά μειοπική ήταν αυτή η προσέγγιση. Χρειάζεται βιώσιμη ανάπτυξη ευρωπαϊκή. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Μέσω του ορισμού του μηχανικού αυτού για τη σύνδεση της Ευρώπης, συνδέοντας στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αλλάξει αποφασιστικά την προσέγγιση μέσω κοινών βάσεων, μέσω εγκασίων τομέων, με μεγάλες δυνατότητες συνέργειας. Γνωρίζουμε όλοι ότι για πετύχουμε τους στόχους της ολοκλήρωσης της αγοράς της ενέργειας και για να φτάσουμε σε μια κοινωνία με χαμηλή εκπομπή οξυδίων του άνθρακος πρέπει να αναπτύξουμε δικτύα και ενεργειακές διασυνδέσεις, διαδικτυώσεις για να εκμεταλλευτούμε και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για να έχουμε επίση να εξασφαλίσουμε και τον ασφαλή εφοδιασμό σε ενέργεια. Εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή όσον αφορά τον τελικό σκόπο, αλλά λείπουν κάποιε λεπτομέρειε όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά του πόρου που διατίθεται. Όπω αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στι 4 Φεβρουαρίου του 2011, το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων θα πρέπει να προέρχεται από την αγορά. Αλλά θα πρέπει να διερωτηθούμε πο... μέχρι το 2020 πόσα θέλει να επενδύσει ο ιδιωτικό τομέα πέρα από τους πόρους που αναφέρονται στην πρόταση για τον ενεργειακό τομέα, βλέπουμε ότι είναι λίγο παραπάνω από 9 δισεκατομμύρια έναντι των εκτιμωμένων 200 δισεκατομμύριων που υπολογίζονται ότι χρειάζονται συνδέσεις και ενεργειακές υποδομές. Ένα εικοστό από το συνολικό ποσό που αιτείται. Ε, συζητούμε αυτή την πρόταση ενώ το πακέτο για τις πολι... πολιτείς δημοσιονομικές προπτικές πρέπει να συζητηθεί χρειάζεται να δημιουργήσουμε μέσα οικονομικά καινοτόμα, όπως είναι τα project bonds, που θα πρέπει να προβλέπουν στοιχείο μόχλευσης για να καλυφθεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των απαιτουμένων και των παρεχομένων. Ε, δεν θέλουμε ε, να υπονομεύσουμε την υλοποίηση των στόχων. Θα πρέπει να εστιαστούμε στις στα διαθετικά ταμεία, τις διάφορες μορφές χρηματοδότησης που έχουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ταμεία για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής, για να εξισορροπηθούν οι μεγάλες επενδύσεις που χρειάζονται ε, μέσω της πρότασης αυτής και που κυρίως αφιερώνονται οι επενδύσεις αυτές που αναφέρονται στην ε, μεταφορά και η κατανομή των διαφόρων, ε, στους διαφόρους τομείς και για την ενέργεια δεν αναφέρεται. Δεν καθόρισε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς οι χρηματοδοτήσεις στα κονδύλια θα διανεμηθούν μεταξύ των διαφόρων έργων κοινή ωφελία και πώς μοιράζονται μεταξύ των τομέων του, της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου πιο συγκεκριμένα. Αυτά ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πυρίλο. Ο κύριος Ντεμπάκα έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που σήμερα προβαίνουμε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην κοινή αυτή συνεδρία των δύο επιτροπών, διότι θεωρώ πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να εξετάσει από κοινού το θέμα αυτό, δηλαδή με πλήρωνες επιτροπές, διότι χρειαζόμαστε μια κοινή θέση, όπως και το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε τη διευκόλυνση αυτή. Χρειάζεται να επενδυθούν πολλά δισεκατομμύρια και, στην, και στις μεταφορές και στις επικοινωνίες και στην ενέργεια. Και βέβαια η διευκόνηση συνδέοντας στην Ευρώπη θα αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για τη χρηματοδότηση. Πρώτα θα κάνουμε συζήτηση για τον πολιετή προπολογισμό και εδώ συμφωνώ με τους προλαλήσοντες ότι οι, οι συζητήσεις αυτές πρέπει να διεξαχθούν σωστά, πρέπει να πρικιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα απαραίτητα κονδύλια ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν που συνεργαζόμαστε. Θεωρώ επίσης σημαντικό τα δημόσια κονδύλια που διαθέτουμε να χρησιμοποιηθούν σωστά και να αποτελέσουν μοχλό για την προσέλκυση και άλλων ιδιωτικών κονδυλίων. Υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα και πολλές ασάφειες στην πρόταση. Χρειαζόμαστε όμως απολύτως την διαφάνεια και τη σαφήνεια για να μην παραμείνουν μακριά οι ιδιωτικοί, οι ιδιώτες μάλλον επενδυτές. Η πιλωτική φάση των προγραμμάτων μπορεί να καταστήσει σαφές και το πώς προτίθεται να προωθήσει το έργο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν τα διάφορα μέρη του προγράμματος. Για, για τον τομέα των μεταφορών είναι σαφές προς τα που θα κατευθυνθούμε. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω και τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Και εδώ νομίζω πρέπει να διατηρήσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Και μια τελευταία παρατήρηση για τι μεταφορέ Είδα ότι στην πρόταση προβλέπονται σημαντικά δημοσιονομικά κονδύλια για την εσωτερική ναυσιπλοεία και για το σιδηρόδρομο. Νομίζω ότι και οι δύο αυτοί φορείς των μεταφορών πρέπει να τύχουν ίσης μεταχείρισης. Ναι. Και τα επιχειρηματικά σχέδια των φορέων πρέπει και αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταλήξουμε σε μια ξεκάθαρη θέση σε συνεργασία των διαφόρων επιτροπών και αν μας επιτύχει τελικά αυτό θα έχουμε μια ξεκάθαρη θέση και θα μπορούμε στην βάση αυτής να συζητήσουμε και με την Κομισιόν και με το Συμβουλίο. Ευχαριστώ. Κύριο Τέρμε, ασκιώδη συγητής των Πρασίνων στην Ήτρα. Για τρία λεπτά, παρακαλώ, κύριε Τέρμε. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, καταπληκτική αυτή η ευκαιρία για συνάντηση και συνεργασία με τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Πολύ σημαντικό το θέμα και πιστεύω ότι ε, η πρόσβαση στο κεφάλαιο είναι το πιο επίγον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το ε, επισήμαναν και οι κύριοι Καντσιάν και Πυρίλο. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό για να βοηθήσουμε ε, την, την, τα προβλήματα, να λυθούν τα προβλήματα στις ε, κεφαλαγορές. Στην ε, Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, ακόμη και αν έχει κάνεις ένα πολύ καλό πρόγραμμα, πηγαίνει στην τράπεζα προσπαθεί να πάρει δάνειο με τη δεδομένη κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ιταλία για παράδειγμα και δεν μπορεί. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την πρόσβαση στο κεφάλαιο αξιοποιώντα αυτά τα κονδύλια του συνδέοντα την Ευρώπη. Εκεί είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όπως είπε και ο Μάικλ, με τις ε, μεταφορές ε, έχουμε περισσότερο ε, δημόσια κονδύλια, ενώ στην ενέργεια ε, ξεκινάμε με κάποια δίκτυα ε, και από ένα σημείο και μετά, μετά από κάποια χρόνια, αναλαμβάνει ιδιωτικό τομέα. Ενώ στι μεταφορέ έχουμε περισσότερο επιχορηγήσει. Στην ενέργεια μα ενδιαφέρει περισσότερο πρόσβαση στο κεφάλαιο. Και αν στη μεταφορά βλέπουμε ότι ε, το ζώο είναι διαφορετικό, οι κανόνε είναι διαφορετικοί. Χρειαζόμαστε όμω κάποιοι γενικοί κανόνε περιβαλλοντική νομοθεσία, πρόοδο κτλ. Αλλά για την ευρυζωνία, την ενέργεια και τις μεταφορές μπορεί οι λεπτομέρειες να είναι διαφορετικές, αλλά το πλαίσιο μπορεί να είναι γενικό. Και έχουμε και το θέμα του παραρτήματος. Μερικοί θέλουν παράρτημα για τις μεταφορές, άλλοι θέλουν παράρτημα για την ενέργεια και αυτό είναι κάπως περίπλοκο. Τελευταία παρατήρηση. Στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστά μόνο μεταφορές ενέργεια και τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, αλλά να έχουμε και κάποια κοινά σχέδια. Θα ήθελα να πω στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι για το PV, τα FE, δίκτυα, ε, EV, από το PV ηλεκτρικό πεδίο και μετά χρειαζόμαστε ε, FE δίκτυα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό όμως σε μια λογική που κατά παράδοση χρησιμοποιούσαμε ξεχωριστούς τρόπους προσέγγισης και κάθε το ήταν ξεχωριστός. Πώς ε, θα μπορέσει ο εκτελεστικός οργανισμός να ε, υιοθετήσει μια πιο οριζόντια προσέγγιση. Το ίδιο θα μπορούσαμε να έχουμε και στις σιδηροδρομικές μεταφορές με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφή και μεταφορές, σιδηροδρόμους να δώσουμε έμφαση όσο το δυνατόν πιο οριζόντια δηλαδή προγράμματα και σχέδια. Κύριο Κράμερ, τρία λεπτά. Νομίζω πρώτα πρέπει να αναλύσουμε γιατί τα τελευταία 20 χρόνια, παρόλο που δαπανήθηκαν πολλά χρήματα, η Ευρώπη δεν ενώθηκε. Πολύ λίγο μόνο. Και αν εξετάσει κανεί τον χάρτη σήμερα, θα διαπιστώσει ότι τα κενά βρίσκονται ακριβώ εκεί, συμπίπτουν δηλαδή με τα σύνορα. Θα ρίξω λοιπόν λίγο νερό στο κρασί μου. Θα πω ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, αλλά μια διαφορετική πολιτική. Διότι αν βάλουμε, αν επιλέξουμε μόνο πολύ λίγα μεγάλα έργα για τα υπόλοιπα που είναι σημαντικά, θα μείνουν στη μέση. Για μένα δεν με ενδιαφέρει εάν το τούνελ του Μπρένερο θα είναι έτοιμο το 2050 κατά 50 ή 60 ή 70%. Εμείς θέλουμε όμως άλλα πράγματα εδώ. Θέλουμε ένωση της Ευρώπης, διασφάλιση της κινητικότητας και επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Εδώ χρειάζονται και μικρά έργα λοιπόν. Παράδειγμα, ο διάδρομος Στοκχόλμη-Παλέρμο. Υπέροχος. Υπάρχει στο μέσον αυτού του διαδρόμου ένα μικρό Erfurt-Niremberg, μόνο γερμανικό. Επ' αυτού έχει δοθεί πολύ χρήμα ευρωπαϊκό, αλλά για το τελευταίο μικρό κομματάκι μέχρι το Μόναχο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο στη Γερμανία, οι χώρες μέλη λένε ε, είναι μεν εθνικό το έργο αλλά έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, παίρνουν τα χρήματα και δεν επενδύουν εκεί που θα έπρεπε, που είναι στα σύνορα, διαμεθοριακά δηλαδή. Αλλά βέβαια δεν υπόσχονται πολλά κέρδη τα διαμεθοριακά έργα. Πολύ περισσότερα υπόσχονται αυτά που βρίσκονται μέσα στο κέντρο των χωρών μελών. Από τους πέντε διαδρόμους μας φτάνει ένας έχουμε τον πράσινο διάδρομο, έχουμε για το, τη, τη μεταφορά του φορτίου από ένα τρόπο μεταφορά σε άλλο. Είναι πολλά, είναι πέντε συνολικά. Βέβαια, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο σε μεγάλα νούμερα, πρέπει να κάνουμε πράξεις στα μικρά. Οι περισσότεροι στην Ευρώπη κινούνται σε ακτίνα λιγότερη των 50 χιλιόμετρων. Σε αυτά πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος λοιπόν. Ένα παράδειγμα. Cross border, πολύ σημαντικό. Αλλά και εκεί πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Τη δήλωση δεν είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό. Για παράδειγμα, λένε οι Σλοβάκοι, Είμαστε τόσο μικρή η χώρα μας που όλες οι διασυνδέσεις με τον σιδηρόδρομο είναι διαμεθοριακές. Πρέπει λοιπόν εκεί να γίνει κάτι. Σήμερα το πρωί τα έλεγα αυτά, ανάμεσα στο Βερολίνο και στην Μπρέσλαου στην Πολωνία. Οι Πολωνοί έχουν κάνει την ηλεκτροκίνηση της, ε, του σιδηροδρόμου μέχρι τα σύνορά τους. Οι Γερμανοί τους μένουν ακόμα 50 χιλιόμετρα. Ναι, δεν πειράζει. Δισεκατομμύρια για το τούνελ του Μπρένερ ε, δεν υπάρχουν χρήματα για εκείνα τα 50 χιλιόμετρα. Με αποτέλεσμα τρομερές καθυστερήσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειαζόμαστε αυτή την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία που σημαίνει ένωση της Ευρώπης. Αυτό δεν θα γίνει με τα μεγάλα έργα. Χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική. Όταν θα την αποκτήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική, τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική των μικρών έργων, τότε θα έχουμε και ε, τα χρήματα και για τα μεγάλα έργα. Ο κύριος Ζήλε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αυτός ο μηχανισμός ε, που προτείνεται ε, είναι πολύ σημαντικός, καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χρειάζεται συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων, υποδομών, μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι κάτι που αφορά όχι μόνο την πτυχή του σχεδιασμού αλλά και τη αμόφωση πολιτικής. Η αρχή της ε, παρόμοιας χρηματοδότησης στην προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη διασύνδεση των περιφερειών της Ευρώπης την ένωσή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μιλάμε για ένωση με κομμάτι του κόσμου. Κάτι που είναι σημαντικό για την Ανατολική Ευρώπη. Σύνδεση με τη Ρωσία, Φερρυπίν. Και την κοινοπολιτεία της Ομοσπονδίας. Πρέπει να δημιουργήσουμε ε, διάφορα έργα που δίνουν προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή. Και είναι σημαντικό να μην χαθεί η προσέγγιση των διαδρόμων διότι γίνονται διάφορες προσπάθειες να παραιτηθούμε από αυτόν τον ορισμό και αυτή την προσέγγιση και σε διαφορα κρατημέλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μην χαθούν τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Συνοχής στο μηχανισμό αυτό για τη σύνδεση της Ευρώπης. Διαφορετικά θα απομείνει μόνο το όριο της χρηματοδότησης που θα αυξηθεί λίγο, 40% του προϋπολογισμού. Και γνωρίζουμε όλοι ότι στις χώρες που χρησιμοποιούν ε, το Ταμείο Συνοχής δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την προσέγγιση. Για τα συνδρομικά έργα πρέπει να πληρώσουμε 70% τα κράτη-μέλη ε, και κανονικά αυτό δεν γίνεται ποτέ στην πράξη. Αν χάσουμε το Ταμείο Συνοχής δεν θα εφαρμοστούν τα έργα των διαδρόμων θέλω να δημιουργήσουμε. Θα υπάρχουν διασυνδέσεις με τρίτες χώρες και όχι με τη Δυτική ή Κεντρική Ευρώπη. Και παρακαλώ να μην χαθεί αυτή η διασύνδεση που είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην χάσουμε τα πάντα. Ακόμα και αν δεν είναι η ιδεώδης λύση, τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Συνοχής είναι ένα σημαντικό ποσό εντός του μέσου αυτού της σηματοδοτικής διευκόλυνσης. Αυτό πρέπει να το αποφύγουν πάση θυσία να χαθούν τα χρήματα. Ευχαριστώ κύριε Ζήλε. Ο κύριος Βιντάλ έχει το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν έχουμε δύο τομείς στους οποίους η οι επενδύσεις ε, έχουν τη μέγιστη απόδοση και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, σίγουρα οι δύο τομείς αυτοί είναι οι υποδομές και η έρευνα στην καινοτομία και στην ανάπτυξη. Έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κανονισμό για τι κατευθυντήρε γραμμές ό,τι αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Έχουμε τον κανονισμό για κατευθυντήρε γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, ανάπτυξη του, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και φυσικά έχουμε και τον ορίζοντα του 2020. Οι τεράστιες προσπάθειες ε, που κάνουμε μεταξύ μας και είναι πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η στενή συνεργασία μεταξύ δύο επιτροπών, Ήτρε και Τράνη, τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουμε για να ενοποιήσουμε κριτήρια, διαδικασίες, για να βελτιστοποιήσουμε ε, τον τρόπο χρηματοδότησης ε, των υποδομών. Όλες αυτές οι τιτάνιες προσπάθειες θα είναι περιτές αν δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κονδύλια για τη χρηματοδότησή τους. Η χρηματοδότηση είναι ο ακρογωνίος λήθος, ε, αλλά και ταυτόχρονα και η λιδία λήθος αυτών των ευρωπαϊκών πολιτικών για τις υποδομές. Γιατί χωρίς χρηματοδότηση τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Η κατάσταση δυστυχώ επιδεινώνεται λόγω της χρηματοπιστωτικής ε, δινής κρίσης που αντιμετωπίζουν περισσότερο ορισμένες χώρες μέλη οι κυβερνήσεις τους ε, υφίστανται τεράστιες πιέσεις προκειμένου να εξηγιάνουν τα οικονομικά τους, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας βρίσκεται με δεμένα χέρια. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν ευρηματικού ε, και καινοτόμου τρόπου για να κινητοποιήσουμε κεφάλαιο, να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στο κεφάλαιο. Από αυτή την άποψη, η πρόταση του κανονισμού που ιδρύει αυτό το μέσο διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτή την άποψη λοιπόν η πρόταση είναι πολύ επίκαιρη και πολύ εύστοχη και αξιέπαινη. Ένα σωστό κριτήριο επιλογής είναι μια ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους. Βέβαια δεν υπάρχει αυτό το κριτήριο για να κρίνουμε την επιλεξιμότητα. Γιατί μερικές φορές ακούμε και το επιχείρημα της ε, ε, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Και αυτό το επιχείρημα έχει το βάρος του ιδιαίτερα όταν μιλούμε για παρέμβαση των κοινοτικών οργάνων. Ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει να δούμε και το θέμα των ενεργειακών νησίδων, αν πραγματικά θέλουμε μια γνήσια ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Η ανάπτυξη των ε, υποδομών ενέργειας και μεταφορών είναι πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταποκρίνεται και στους ε, ιδρυτικούς της ε, στόχους. Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουμε ε, για να εξασφαλίσουμε αυτή την χρηματοδότηση που επικρίνεται πολλές φορές τριμήτατα εξαιτίας της ε, αδιαφάνειάς της. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού, αυτού του μέσου διευκόλυνσης για το, το συνδέοντα στην Ευρώπη και η ανέβρεση και ενοποίηση κριτηρίων για την χρηματοδότηση των διαφόρων υποδομών είναι σημαντικό βήμα προόδου. Ευχαριστώ. Τρία λεπτά Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ήδη λέχθηκαν από τους συναδέλφους μου και έτσι και αλλιώς και στο Κοινοβούλιο έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Προετών, θυμάστε, μας είχαν δείξει αυτούς τους θαυμάσιους χάρτες που σημείωναν όλα αυτά τα έργα από τα οποία πολύ λίγα τελικά υλοποιήθηκαν. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε τρία πράγματα. Πρώτα, χρειαζόμαστε το ταμείο αυτό να έχει λεφτά. Η δεμή όλα είναι κενές υποσχέσεις. Είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόταση της Επιτροπής που προβλέπει 31,7 δισεκατομμύρια. Είναι περισσότερο από αυτά τα 8 δισεκατομμύρια που έχουμε στην, ε, στον προϋπολογισμό των TEN-T. Πρόκειται όμως για το κύριο δίκτυο και μόνο γι' αυτό χρειαζόμαστε 500 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για ένα ποσό που με κάποιο τρόπο πρέπει να συλλεχθεί μέχρι το 2030. Με αυτά τα 31,7 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα σε αυτά ε, υπάρχουν και κονδύλια που έχουν προέλθει από καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς ίσως προέλθουν και άλλα κονδύλια. Αλλά δεν μπορεί να περιμένει κανείς πάρα πολλά πράγματα, διότι ίσως γίνει η κατάσταση ακόμα περιπλοκότερη με την αναζήτηση αυτών των κονδυλίων και ίσως και τελικά να μην και καλύτερη χρηματοδότηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που θα προέλθουν υποτίθεται από το Ταμείο Συνοχής. Θα πρέπει βέβαια να περιμένουμε πολύ έντονη αντίδραση από το Συμβούλιο Υπουργών και κυρίως από ορισμένες βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να κάνουμε κάθε το δυνατό για να τις καθησυχάσουμε τις χώρες αυτές, χωρίς βέβαια να χάσουμε από τα μάτια τον γενικότερο στόχο και κυρίως τις γενικότερες αρχές να καθησυχάσουμε το Συμβούλιο δηλαδή ότι τα κονδύλια άνα ενδιαφερόμενη χώρα θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα και να κατορθώσουμε η χρηματοδοτική ικανότητα των χωρών να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά. Δεύτερο, να συμφωνήσουμε στο πού θέλουμε να συγκεντρώσουμε τις προσπαθίες μας. Έργα δηλαδή τα οποία προσφέρουν πραγματική, γνήσια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και βέβαια αυτά να ταιριάζουν και με τους βασικούς μας εσωτερικούς στόχους περιλάβαμε στη Λευκή Βίβλο. Είπαμε ότι επιζητούμε βιωσιμότητα στις μεταφορές, εσωτερικές ε, υδάτινες μεταφορές, σιδηρόδρομο κλπ. Ένα τρίτο θέμα που πρέπει να μην είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα που δεν μπορούν να μείνουν χωριστά από τη συζήτηση που γίνεται τώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες άσκησης επιρροής από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση των έργων. Χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες να δίνουμε τις κατευθύνσεις, καθώς επίσης και τεχνική διαλειτουργικότητα. Πρέπει να διασυνδεθούν οι ευρωπαϊκές αυτές επιχορηγήσεις με ορισμένους όρους και να φροντίσουμε ακόμη ώστε τα κονδύλια να διατίθενται με τρόπο αποδοτικό, διότι ο στόχος είναι μέσα από τα δίκτυα αυτά να ενισχυθεί και να ανδρωθεί η ενιαία αγορά. Άρα χρειάζονται ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν, αλλά νομίζω ότι αν επιδιώξουμε ενωμένοι τους στόχους αυτούς, θα τα καταφέρουμε. Ο κύριος Γκρός για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζουμε με ποιον θα συνομιλήσουμε αύριο, στο μέλλον δηλαδή, το Συμβούλιο και να κάνουμε προσπάθεια κοινή για να τους πείσουμε. Να μην προκύψει ανταγωνισμός μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η πρόταση είναι νέα και είναι καλή. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν και αυτοί που δεν είναι μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Όπως είπε ο κ. Σελκαντράουι, γνωρίζουμε και από πριν ότι αν προσθεθούν απλώς διάφορες εθνικές προτεραιότητες, δεν φτάνει αυτό για να φτάσουμε σε ένα δίκτυο ευρύ ευρωπαϊκό που θα αποκαταστήσει την διασύνδεση και με τις περιφέρειες. Πρέπει να διδαχθούμε από το παρελθόν και να αποφύγουμε να προσπαθήσουμε να περιλάβουμε και το τελευταίο μικρό εργάκι στους καταλόγους αυτούς. Πρέπει να τα εξηγήσουμε αυτά και στο Συμβούλιο και στις χώρες και στις περιφέρειες. Το δεύτερο είναι να βάλουμε κέντρα βάρους. Είπε προηγουμένως κάποιος οι διαμεθοριακές συνδέσεις. δεν ωφελείται τότε μία από τις δύο χώρες, ωφελούνται και οι δύο. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ε, θέσπιση προτεραιοτήτων. Και γι' αυτό πρέπει να τεθεί το Συμβούλιο ενώπιον των ευθυνών του. Και να του ρωτήσουμε, θέλετε, θέλει η συγκεκριμένη χώρα να είναι μέλος του δικτύου ή θέλει να μείνει απ' έξω. Θέλετε να αποκλείσετε το δίκτυο που θέλετε να φτιάξετε από άλλες χώρες ή θέλετε να συνεργαστείτε διαμεθοριακά. Πρέπει να τους πούμε λοιπόν καθαρά ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα θαυμάσιο εργαλείο που φτάνει μέχρι και τις ακραίες περιφέρειες. Περιλαμβάνει και τους βασικούς κανόνες της Λευκής Βίβλου και για, του, και για τους διάφορους τρόπους μεταφορών. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε διαφορετική βάση τίσως με το Συμβούλιο. Και σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά πρέπει να πούμε επίσης καθαρά και εδώ απευθύνομαι λίγο και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών Αυτά που προτείνονται εδώ είναι το ελάχιστο, διότι αυτά που προτείνονται εδώ συνολικά είναι λιγότερα από προηγουμένως, από παλαιότερα. Είχαμε ζητήσει παλαιότερα 60 δισεκατομμύρια και μας έδωσαν 8. Τώρα λέμε 20 συν 10 από το Ταμείο Συνοχής, συν 10 για την ενέργεια και για τις επικοινωνίες. Όχι, δεν πάει έτσι. Και στο Περιφερειακό Ταμείο έχουμε πάνω από 80 δισεκατομμύρια επενδύσει για την κινητικότητα. Και τώρα έχουμε φτάσει μάλιστα να λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε ορισμένε περιφέρειε δεν μπορούν να γίνουν πλέον επενδύσει για την κινητικότητα. Πρέπει να πούμε λοιπόν στην Επιτροπή Προπολογισμών ότι αυτά που προβλέπονται εδώ είναι το ελάχιστο, είναι το μίνιμουμ. Και, για να και πρέπει να είμαστε συνεπεί ώστε οι επενδύσει αυτέ να είναι συν για όλε τι χώρε. Και σε περιόδους εξοικονομήσεων είναι απαραίτητο να γίνουν επενδύσεις για την βελτίωση των περιφερειών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και τα υπόλοιπα γραπτός. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κουμουτσάκος για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν θα χρησιμοποιήσω τα τρία λεπτά γιατί δεν έχω πολλά να προσθέσω μετά την τόσο ξεκάθαρη τοποθέτηση του Ματιέ Γκρός. Ε, <clears throat> ο στρατηγικός μας στόχος ως Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ακριβώς που αυτό το οποίο μόλις ακούστηκε. Η ευρωπαϊκή επιτυχία των διευρωπαϊκών δικτύων. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια λογική αθρίσματος εθνικών προσπαθειών, αλλά μια συνολικής και συλλογικής προσέγγισης σε ένα τόσο μεγάλο θέμα. Βεβαίως, το SEF, το Connecting Europe Facility, είναι ένα νέο εργαλείο. Είναι ένα θετικό εργαλείο και πρέπει να είναι στόχος μας να το διατηρήσουμε και αν είναι δυνατόν να το βελτιώσουμε. Ο ρεαλισμός λέει ότι πρώτος μας στόχος είναι να το διατηρήσουμε. Βεβαίως η διαπραγμάτευση και κανείς δεν έχει ψευδεστήσεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και πάρα πολύ πολύπλοκη. Σε τουλάχιστον δύο αλληλεξαρτώμενα επίπεδα. Το επίπεδο των, του πολιετούς οικονομικού πλαισίου και μετά το επίπεδο του ΣΕΦ. Ως ε, ένας από τους δύο εισηγητές του κανονισμού για τις κατευθυντήριες γραμμές των διευρωπαϊκών δικτύων, πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλο προβληματισμό και ανησυχία, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, η πορεία των διαπραγματεύσεων και για το πολιετές οικονομικό πλαίσιο και για το ΣΕΦ επηρεάζει άμεσα και την πορεία του κανονισμού για τις κατευθυντηρίες γραμμές. Οφείλουμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Αν θα υπάρχουν αριθμοί, αν θα υπάρχουν νούμερα, αν θα υπάρχουν κονδύλια, δεν θα υπάρχουν. Η λογική και η ευελιξία λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια. Ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, διότι αν ζητήσουμε να υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά, αυτό θα καθυστερήσει πάρα πολύ διαδικασία. Πάντω, καμία από τι δύο σχολέ σκέψη δεν είναι πανάκια, δεν είναι το πρόβλημα. Αλλά σίγουρα η ευελιξία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καλύτερη. Και ένα τελευταίο σημείο, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πραγματικά να ξέρω, επειδή ο ιδιωτικό τομέα πρόκειται να παίξει και, εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να παίξει σοβαρό επενδυτικό ρόλο, πώ αντιλαμβάνεται ο ιδιωτικό τομέα το ΣΕΦ. Το θεωρεί ένα θελκτικό εργαλείο. Τους, τους τραβάει. Το θεωρούν ότι μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις ή το βλέπουν με επιφυλακτικότητα ή ακόμα χειρότερο με άρνηση. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο εάν θα μπορούσαμε σε αυτή τη ζήτηση να το ξέρουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε τρία λεπτά κύριος Μπράντμπερν. Ευχαριστώ. Δεν θα χρειαστώ καν. Ε, έχουμε το φάσμα, αισθάνομαι σαν να είμαστε στο φάσμα του συμποσίου. Από αυτό που ακούσαμε μέχρι στιγμής από τη συζήτηση, διαπιστώνουμε ότι επικρατεί ένα κλίμα εφορία. Τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα νέα μέσα, όλε αυτέ τι νέε διευκολύνσει και ούτω καθεξή. Χθε θα θυμάστε ότι στην ε, συνεδρίαση ανέφερα κάποια σχόλια για τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα, για τι χρηματοπιστωτικέ πτυχέ, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα των ομολόγων ε, έργου και δεν έλαβα ικανοποιητικέ απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να τα παραλάβω για να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι τη Σύτρε τι γίνεται με τις ευθύνες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά ε, τα ομόλογα έργου. Ποιος ε, θα επιτηρεί, ποιος θα επιβλέπει τον τρόπο εφαρμογής αυτών των μέσων και αυτών των διευκολύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομίζω ότι έχει την εμπειρογνωμοσύνη για να εξασφαλίσει τέτοια επιτήρηση επίβλεψη, αλλά ούτε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχουν προβλήματα, λοιπόν, σοβαρά προβλήματα διακυβέρνηση για τι χρηματοπιστωτικέ πτυχέ αυτή τη πρόταση και χρειαζόμαστε κάποια διαφάνεια για το πώ θα εφαρμοστεί, πώ θα λειτουργήσει αυτή η διακυβέρνηση και για τα ίδια τα μέσα αυτά τα χρηματοδοτικά, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο του μέσου αυτού του συνδέατο στην Ευρώπη, του ΣΕΦ. Επίσης υπάρχει και θέμα δομής. Τι δομή θα έχει αυτό το νέο δημιούργημα, αυτό το νέο χρηματοδοτικό μέσο. Στο παρελθόν ασχολήθηκα με προγράμματα διευρωπαϊκών δικτύων και όλοι λέμε τι ωραία που είναι όλα αυτά, είμαστε ενθουσιασμένοι και διεκδικούμε όλο και περισσότερα κονδύλια, αλλά έχουμε την ε, στιγμή χρηματοπιστωτική πραγματικότητα διεθνώς. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ ελαστικοί στην προσέγγισή μας. Κάποιες χώρες της Ένωσης και κάποια τμήματα της Ένωσης θα επιμείνουν ιδιαίτερα στους διαδρόμους τους συνδέοντας την Ευρώπη. Άλλοι θα επιδιώξουν άλλες δραστηριότητε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ αναφέρθηκε στην αποσυμφόρηση των στενοπών. Αυτό είναι ένα θέμα που γρήγορα θα είναι αποδοτικό και θα αποφέρει καρπού στη χρήση των κονδύλιων του συνδέοντας στην Ευρώπη. Τέτοιου είδους προσέγγιση χρειαζόμαστε, ελαστική και όχι μία άκαμπτη και προκαθορισμένη προσέγγιση που θα είναι τελείως αδιάλακτη και θα μας φέρει ε, στην κατάσταση που είμαστε σήμερα με τα διευρωπαϊκά, γιατί ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Γι' αυτό και οι καλές προθέσεις και του μέσου αυτού μπορεί να μας οδηγήσουν στην κόλαση κάποια στιγμή προσοχή λοιπόν. κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω στην συνεδρίασή μας τους εκπροσώπους της Επιτροπής Ήτρε, τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση Τραν και Ήτρε. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας είναι θέματα κοινού ενδιαφέροντος, γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε με τι κριτήρια θα προσδιορίσουμε τα προγράμματα και σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. Σε ό,τι αφορά τα 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Συνοχής που θα αφιερωθούν στην ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών των χωρών που πληρούν τα κριτήρια της συνοχής. Χρειάζεται μια εθνική κατανομή αυτών των 10 δισεκατομμύριων. Και έχω μια ερώτηση και προς τους συνεισηγητές και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 11, εδάφιο 2 του κανονισμού για την διευκόλυνση αυτή του συνδέοντας στην Ευρώπη. Αναφέρεται εκεί ότι οι εφαρμοστεί κανόνες για τον τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο του κανονισμού θα ισχύσουν για συγκεκριμένους διαδρόμους και θα χρηματοδοτηθούν από τα 10 δισεκατομμύρια. Κάπου αλλού αναφέρεται ότι ε, για τέτοιου είδους προτάσεις θα δοθεί προτεραιότητα στα σχέδια και προγράμματα που πληρούν τις εθνικές προτεραιότητες ε, για τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής. Μιλούμε δηλαδή για προγράμματα που τηρούν τους εθνικούς όρους κατανομής των κονδυλίων. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στο άρθρο 9 σημείο 6 αναφέρονται τα ετήσια προγράμματα και τα πολιτικά προγράμματα που θα εγκαινιαστούν μετά από προκήρυξη διαγωνισμών. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι αυτά τα ετήσια και πολιτικά προγράμματα θα μπορούν να περιλαμβάνουν επιπλέον κανόνες για την υποβολή προτάσεων και διαγωνισμών. Θα ήθελα να περιοριστούμε στα κριτήρια του κανονισμού και να μην προσθέτουμε νέα κριτήρια. Εκτός και είναι μόνο διαδικαστικά και αν δεν αλλάζουν την ουσία του κανονισμού. Θα ήθελα και πάλι να αναφερθώ σε αυτά 10 δισεκατομμύρια του Ταμείου Συνοχής. Και έχω και μία ακόμη ερώτηση προς την Κομισιόν. Αναφέρεται η, η συγκεντρωτική ε, ε, διαχείριση αυτών των κονδυλίων ίσως μέσω ενός ε, εκτελεστικού οργανισμού. Εδώ όμως έχουμε αντίφαση με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου Συνοχής. Επίσης σας παραπέμπω στο κεφάλαιο της ενέργειας και για το φυσικό αέριο και για τον ηλεκτρισμό. Μιλήσαμε για 12 κατά προτεραιότητα διαδρόμους και υποβάλλονται διάφορα κριτήρια και διατάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οι απαιτήσει των αγορών, τιμή των καυσίμων, δυνατότητα αποθήκευσης και στην περίπτωση των μεταφορών οι περιφέρειες είναι αυτές που θα πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια. Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες της πληροφορικής και της ε, επικοινωνίας. Θα δώσουμε έμφαση στην ε, ευρυζωνία και στις ψηφιακές ε, πανευρωπαϊκές υπηρεσίες. Ποιες είναι οι υπηρεσίες ε, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα πρέπει να παρέχονται διασυνοριακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, ε, τα θέματα της ε, ανάπτυξης των επικοινωνιακών δικτύων και των νέων και των παλιών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη. κυρία Σέναλοβα, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι γενικώ η ιδέα για το χρηματοδοτικό μέσο συνδέοντας την Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία, κρίσιμη θα έλεγα, για την εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε καλύτερες διασυνδέσεις στην Ευρώπη, κάτι που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Παραμένουν όμως πολλά ακρεμή ζητήματα ακόμη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΣΕΦ, το μέσο αυτό συνδέοντας στην Ευρώπη, ε, και το, τη σχέση του με το Ταμείο Συνοχής. Τι γίνεται με προγράμματα που δεν θα κρυθούν επιλέξιμα με βάση το ΣΕΦ. Θα μπορούσαν παρόλα αυτά τα προγράμματα αυτά να τύχουν χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Μία άλλη ερώτηση μου αφορά τη δυνατότητα καλύτερου συντονισμού. Δεν ξέρω αν θα βελτιώσουμε τον συντονισμό μας με μεγαλύτερη συγκέντρωση της διαχείρισης. Χρειαζόμαστε πάντως καλύτερο συντονισμό, ιδιαίτερα για τις διασυνοριακές διασυνδέσεις. Αλλά δεν ξέρω αν ο συγκεντρωτικός τρόπος διαχείρισης είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε αυτόν τον καλύτερο συντονισμό. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι η εδαφική συνοχή και η αλληλεγγύη. Όχι μόνο επειδή αναφέρονται και στη Λευκή Βίβλο, αλλά γιατί χρειαζόμαστε συνέργεια των επενδύσεων και αποτελεσματική χρήση των, και αξιοποίηση των πόρων. Και επίση τα 10 δισεκατομμύρια ταμείου συνοχή, άλλο σημαντικό ζήτημα. Κυρία Μπιλβά Κύριε Πρόεδρε, με την απεσιοδοξία ποτέ δεν ε, λύσαμε κανένα πρόβλημα. Συμφωνώ με τον κύριο Γκρός ότι έχουμε προβλήματα χρηματοδότηση παντού, αλλά βρισκόμαστε εδώ ακριβώ για να υποβάλουμε προτάσει και να ξεπεράσουμε τι δυσκολίε, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε κάποια στιγμή και λύσει. Εγώ συμμερίζομαι του στόχου ε, του κανονισμού, γιατί πιστεύω ότι όντω θα ε, διευκολύνει τη χρηματοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων και επίσης θα μας επιτρέπει να ελέγξουμε ε, σωστή και έγκυρη ε, διαχείριση και εφαρμογή των προγραμμάτων και με αξιοποίηση των κονδύλιων αυτών από τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι ο κανονισμός αυτός είναι από τα πιο σημαντικά ε, νομοθετικά κείμενα, γιατί επιτέλους το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισαν την ανάγκη για μια κοινή δομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη χώρα των Βάσκων, στα τέλη της δεκαετίας του 80, είχαμε 25 με 30% ανεργία σε ορισμένες περιοχές. Τότε είχαμε περικοπές και ακόμη μεγαλύτερη κρίση. Περικοπές στον προπολογισμό και ακόμη πιο σημαντική κρίση. Και παρόλα αυτά δώσαμε έμφαση στις υποδομές, στην καινοτομία, στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού κλάδου. Γιατί σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει την λιτότητα να τη συνδυάσουμε με μια οικονομική ανάπτυξη ανάκαμψη. Και έτσι καταφέραμε το 2009 να μειώσουμε αισθητά την ανεργία. Θα πρέπει λοιπόν με αυτό το μηχανισμό να υιοθετήσουμε παρόμοια πρότυπα. Να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση παρά την λιτότητα και την κρίση. Σύμφωνα με την ανάγκη για συνοχή, για αντιμετώπιση των διασυνοριακών προβλημάτων ώστε να καταλήξουμε σε μια ανταγωνιστική οικονομία και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και πιστεύω ότι με τα πιλωτικά προγράμματα μπορούμε να έχουμε αίσια αποτελέσματα. Και μάλιστα, εφόσον είναι θετικά τα αποτελέσματα των πιλωτικών προγραμμάτων, μπορεί να προσελκύσουν και ιδιωτικά κεφάλαια. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν που θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί από αυτή την άποψη θέλουμε κάποιες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς εφαρμόζονται και λειτουργούν τα πιλωτικά προγράμματα. Όντως, θα υπάρξουν διαμάχες μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα για το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά το ζήτημα για μας δεν είναι τόσο οικονομικό και χρηματοδότησης. Είναι θέμα πολιτικό, πολιτική συνοτροπίας των θεσμικών οργάνων. Θα καταφέρουμε να αντιληφθούμε τι είναι πρωταρχική σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ποιε είναι οι προτεραιότητες μας και ποιοι οι στόχοι μας. Η χρηματοπιστωτική κρίση θα πρέπει να περάσει σε δεύτερο πλάνο. Θα πρέπει πρώτα να δώσουμε μια λύση στην πολιτική κρίση που αντιμετωπίζουμε. Για δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να ορίσει από κοινού με τα κράτη-μέλη τα κατά προτεραιότητα δίκτυα και να αναλάβει δέσμευση για εξασφάλιση χρηματοδότηση αυτών των πρωτοβουλειών. Στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, έρωτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπήρξαν κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις των κρατών μελών. Χθες ε, συναντήσαμε εδώ τέσσερις ε, νικητές του διαγωνισμού τη ευφυού κινητικότητα, πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ρωτήσαμε από του ε, βραβευθέντε τι περιμένουν από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, μα απάντησαν αυτό που περιμένουν είναι εναρμόνιση και ομοιόμορφε ε, τεχνολογικέ προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι, είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριο Μαρινέσκου για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στις μεταφορές. Έχουμε μία σειρά διαδρόμων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού. Πώς καθορίστηκαν οι προτεραιότητες αυτές. Φαντάζομαι με βάση τις προηγούμενες προτεραιότητες των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Και φαντάζομαι ως προϋπόθεση αναφέρεται το να περνάνε από τις 27 χώρες μέλη. Βέβαια δεν αναφέρεται οικονομική ανάπτυξη. Οι διάδρομοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των σχεδίων και προγραμμάτων. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε το όποιος πρόλαβε ως αρχή. Αλλά στο άρθρο 5 μιλούμε για την ε, γεωγραφική και εδαφική διαφοροποίηση και την εξασφάλιση γεωγραφικής ισορροπίας. Αν συνεχίσουμε με την προσέγγιση αυτή, μέχρι το 2020 δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί κανένας διάδραμος και θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση μετά από 8 χρόνια. Δεν νομίζω ότι ούτε για τον τίτλο δεν θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Το συνδέοντα στην Ευρώπη. Δεν πρόκειται ούτε καν τον τίτλο να υλοποιήσουμε. Θα πρέπει να βρούμε μια διαφορετική λύση. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Και στα θέματα της ενέργειας έχουμε πολλές και διάφορες προτεραιότητες. Και είναι αλήθεια ότι η διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων μεταξύ των κρατών μελών είναι προτεραιότητα, γιατί τέτοια διασύνδεση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Πάντως, η ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και ασφάλεια των ενεργειακών πηγών. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας και εκεί θα πρέπει να αφιερώσουμε τα ισχυρά κονδύλια που έχουμε για να μην διονυστεί αυτή η εξάρτησή μας από μία και μόνο πηγή ενέργειας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία, η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ένα λεπτάκι μόνο, κύριε Πρόεδρε, για να σα υπενθυμίσω ότι μία από τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, η εδαφική συνοχή. Και την περασμένη εβδομάδα ε, η κυβέρνηση της Ισπανίας προσπάθησε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθωθούν κάποια προβλήματα που εντοπίσαμε. Δεν πιστεύετε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σχεδιασμού ε, διαδρόμου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την διάθρωση όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η δική μου περιφέρεια μένει εκτός ε, των σιδηροδρομικών δικτύων και των αεροπορικών δικτύων. Και μόνο τελευταία στιγμή η προηγούμενη Ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να βγάλει την Ριόχα από οποιοδήποτε διασύνδεση δηλαδή στερούμε από μια ευρωπαϊκή περιφέρεια που μέχρι στιγμής είχε καταπληκτική αποτελεσματικότητα στη χρήση των κυρωτικών κονδυλίων και προγραμμάτων, ε, τη στερούμε από τη δυνατότητα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διασύνδεση. Δεν είναι αντιφατικό με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ε, ε, δαφική συνοχή να αφήνουμε εκτός νυμφώνος από τη διασύνδεση, δηλαδή μια ευρωπαϊκή περιφέρεια. Τελευταία στιγμή διόρθωσε η Ισπανική κυβέρνηση τις τάσεις της και αποφάσισε τελικά να συμπεριλάβει και τη Ριόχα στα προγράμματα αυτά και στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποθέτω τώρα ότι ο κ. Πακέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο. Κύριο Πακέ, έχει το λόγο. Τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν επιτρέπει ο χρόνο να καλύψω τι ερωτήσει. Θα σχολιάσω σύμφωνα. Κύριε Πακέ, είμαι σίγουρο ότι ο χρόνο σα επιτρέψει να καλύψετε όλε τι ερωτήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ήτρε και τους ηγητές για αυτή τη συνεδρίαση. Νομίζω ότι δίνει τη σωστή βάση για να ξεκινήσουμε την επεξεργασία αυτού του σημαντικού εργαλείου τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Βασικό στόχο να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη τη Ευρώπη επενδύοντα ε, σε δίκτυα και σωστή τομεί, ε, μεταφορέ, ενέργεια ε, και ηλεκτρονικά και θέλουμε να υπάρχει βιώσιμη κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα. Και όπως πολύ είπατε, η ανταγωνιστικότητα ε, τη ευρεία ενία για πιο εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, αλλά και για καλύτερη ανταγωνιστικότητα για τους τομείς μας, τους, ε, στους οποίους ηγούμεθα το μέσο αυτό αφορά περισσότερο την αποδοτικότητα, την απόδοση και τις ε, συμπράξεις μεταξύ των τριών τομέων, τις συνέργειες μεταξύ των τριών τομέων. Ίσως χρειαζόμαστε και έργα και προγράμματα που καλύπτουν και τους τρεις τομείς. Και θέλουμε συστήματα καθαρών μεταφορών. Θα έχουμε καθαρή ενέργεια έτσι, με τις σωστές υποδομές δικτύωσης και με σταθμούς ε, εφοδιασμούς ενέργεια σε βασικούς κόμβους. Οπότε ε, είναι ένας τομέας που πρέπει να διερευνηθεί. Η πρόταση αφορά τους τρεις τομείς. Κοινά έργα και στους τρεις τομείς. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Το είπαν αρκετά μέλη αυτό. τα τελευταία 5-10 χρόνια με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ενέργεια και μεταφορές επίσης, είδαμε ότι οι επενδύσεις πρέπει να αφορούν την ανάμειξη ιδιωτικών και δημοσίων πόρων. Και πρέπει να βρεθεί και σωστή ισορροπία. Περί αυτού πρόκειται η πρόταση. Ο ιδιωτικό τομέα καλύπτει τι περισσότερε επενδύσει και να δούμε και πού οι δημόσιε επενδύσει είναι αναγκαίε. Τρίτο, πρέπει να βρούμε και τη σωστή διαχωριστική γραμμή. Τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη και οι επιχειρήσεις να φάει επενδύσεις και πού κινείται η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και τα ευρωπαϊκά μέσα για την καινοτομία. Και κάτι άλλο ακούστηκε από πολλούς ομιλητές, σημαντικότατο, που περιέχεται στην πρόταση. Σχέσεις, σχέση μεταξύ αυτής της διευκόλυνσης συνδέοντας στην Ευρώπη και των άλλων μέσων που έχει η Ευρώπη Περιφερειακή πολιτική. Αναφερθήκατε πολύ στα 10 δις που δίνονται για τις χώρες συνοχής όσον αφορά το μέσο διευκόλυνσης για να ωφεληθούν από το ποσοστά συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής. Τα 10 δισεκατομμύρια θα τα διαχειριστούμε όπως οι άλλες συνιστώσεις του ΣΕΦ. Και ζητήθηκαν προτάσεις για να έχουμε μπροστά μας τελικά προγράμματα τα οποία είναι όριμα, αποδοτικά και θα πρέπει να γίνεται σωστή αξιολόγηση ε, ούτω ώστε τα καλύτερα προγράμματα να παίρνουν τα χρήματα και να έχουμε την υψηλότερη ε, προστιθέμενη άξια. Έχουμε βάλει ένα χρονικό όριο του 2020. Έχουμε καινοτομία, έρευνα, ανάπτυξη, όλα αυτά μαζί θέλουμε να εφαρμοστούν και όλα αυτά έχουν ε, διασυνδέσεις μεταξύ τους εν ώψη του 2020 και το μέσο διευκόλυνση της συνδέσης της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνει πολλή δουλειά και εδώ έχουμε και τα project bonds στην πιλωτική φάση και, και το μέσο που συζητάμε επίσης έχει μεγάλη σημασία για τη σύνδεση της Ευρώπης. Τα σημαντικά μέσα χρηματοδότησης θα διευκολύνουν την ιδιωτική χρηματοδότηση και θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα αμόχλευσης και σχετικές επενδύσεις. Και όλοι ανέφεραν κάποια σχέση που υπάρχει μεταξύ του ρυθμιστικού πλαισίου, κατευθυντηρίων γραμμών και του πλαισίου στην ενέργεια και στις μεταφορές που παρέχουν ένα πραγματικό πλαίσιο για την πολιτική και ρυθμιστικό πλαίσιο για να βοηθηθεί η υλοποίηση των έργων όλων των φορέων. Να εντοπιστούν τα έργα αυτά και προγράμματα που δίνουν πραγματικά μεγάλη προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Είναι φιλόδοξη η πρόταση από πολλές πλευρές και από πλευρά κονδυλίων. 50 δις είναι σημαντικό ποσό στα πλαίσια του πολιτού πλαισίου. Δύσκολε είναι οι συζητήσει, διότι υπάρχουν μεγάλε φιλοδοξίε. Το ποσό όμω αυτό ταιριάζει πολύ με τα προγράμματα που εντοπίστηκαν στα παραρτήματα για το μέσο διευκόλυνση ιδιότητα στην Ευρώπη. Έκανε πολλές προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει σχέση μεταξύ των πλαισίων πολιτικών, του καταλόγου των προγραμμάτων και των έργων και των ποσών χρηματοδοτήσεως που θεωρούνται αναγκαία. Έτσι, μέχρι το 2020 θα κινηθούμε για την ολοκλήρωση των δικτύων. Φιλοδοξία όσον αφορά τον προπολογισμό, είμαστε φιλόδοξοι όσον αφορά τι επιλογέ και τη συγκέντρωση και αρκετά φιλόδοξοι όσον αφορά τα μέσα που θα είναι διαθέσιμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία με όλου του ενδιαφερομένους και θέλουμε να σας βοηθήσουμε να προχωρήσετε στην ανάλυση του θέματος. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Οι τρεις εισηγητές έχουν κάτι άλλο, θέλουν να προσθέσουν κάτι. Κυρία Βαλέ, θέλετε να πείτε κάτι βάσει των όσων υπόθηκαν και αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίστε, είχε το λόγο. Μερικά λόγια να πω. Ε, ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν στην συζήτηση, λέει η κυρία Βαλεάν. Και θα συνεχιστεί ο προβληματισμός επί του θέματος και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση και στο καλύτερο δυνατό πλαίσιο. Ο κύριος Ρίκε, κύριε Πρόεδρε, να πω και ε, άκουσα από τη συζήτηση ότι πολύ μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει την αρχή που προτείνεται. Εκφράστηκαν και κάποιες ανησυχίες βέβαια και δυσκολίες που ε, πρέπει να ξεπεράσουμε για να καταλήξουμε τελικά σε ένα καλό κείμενο. Η κυρία Αγιάλα. Και εγώ κύριε Πρόεδρε ήθελα μόνο να πω ότι συμφωνώ με αυτό το τελευταίο και ότι θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε στις βέλτιστες δυνατές λύσεις και εκτός από τη σημερινή συνάντηση θα γίνει και ένα σεμινάριο με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων όπου θα συζητηθούν θέματα τα οποία τέθηκαν σήμερα θα εξετάσουμε και όλα τα έγγραφα που είναι σχετικά με το θέμα και η συζήτηση για το, ότι διευκόλυνση αυτή θα συνεχιστεί. Ο Γιώραν Φάρμ. Ένα σύντομο σχόλιο προς την κατεύθυνση του κυρίου Γκρός ο οποίος έθιξε το θέμα του επίπεδου χρηματοδοτήσεως της διευκόλυνσης και είπε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το ελάχιστον. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Ίσως μάλιστα και η Επιτροπή Προϋπολογισμών μπορώ να πω ότι συμφωνεί. Το πρόβλημα βέβαια είναι οι χώρες μέλη και η κατάστασή τους και το Συμβούλιο. Μην λησμονείτε, η ιδανική προεδρία, η ιδανική κυβέρνηση που έχει την προεδρία δηλαδή, που ασκεί την προεδρία, πολλά πρωτοσέλιδα στον δανεικό τύπο, διότι η δανεική κυβέρνηση ζήτησε εντολή από τη δανεική Βουλή για να μειώσει σημαντικά τα κονδύλια για τη διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Άρα δεν αρκεί η συζήτηση εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στι κυβερνήσει, διότι αλλιώ διακινδυνεύουμε μεγάλε περικοπέ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η πρόεδρος κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είδαμε ότι η συζήτηση ήταν πλουσιότατη. Έβριθε παρεμβάσεων σημαντικών. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Σίμψον για την φιλοξενία του που προσέφερε σήμερα στη συνάντησή μας με την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για τη συνεργασία και σας προσκαλώ όλους στις 24 Απριλίου σε μια συνάντηση, σε ένα δημόσιο σεμινάριο που πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει και θα συμπληρώσει αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι 24 Απριλίου είναι το σεμινάριο που η Επιτροπή Μεταφορών θα είναι φιλοξενούμενη από την Επιτροπή Ήτρε. Χρησιμότατη σημερινή συζήτηση και οι δύο επιτροπές μπόρεσαν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να προβάλλουν επιχειρήματα. Μας περιμένει πολλή δουλειά, όπως είπε ο κ. Φάρμ και άλλοι. Ξεκινήσαμε καλά σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη και των δύο επιτροπών, ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε που ήρθαν εδώ, σε εμά σήμερα και προσβλέπω στις 24 Απριλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ λίγη αυτό το τμήμα συνεδριάσεως. Τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, μην τολμήσετε να φύγετε, πρέπει να συνεχίσετε. Λοιπόν, να μείνετε στι. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Five minutes, colleagues, five minutes. We'll start. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Okay, Ελάτε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη είναι ανακοινώσει του Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών οι οποίοι συντονιστές αποφάσισαν ότι δεν αναλαμβάνεται δράση για, τις, για πέντε έγγραφα έκθεση της Κομισιόν για το Προμασάφα, ΣΑΦΑ. Δεύτερο, βιώσιμοι τρόποι μεταφορών. Η απόφαση εδώ ήταν να ληφθεί υπόψη στην επόμενη έκθεση για την βιώσιμη κινητικότητα και τον τουρισμό. Έγγραφο εργασίας για την ευρωπαϊκή τυποποίηση και το πρόγραμμα δράσης, πάλι no action, ανακοίνωση της Κομισιόν για αποκατάσταση εμπιστοσύνη με βελτίωση της συνεργασίας και η Γενική Έκθεση για τις δραστηριότητες της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011, πάλι εδώ, no action. Για το ΣΤΟΑ η απόφαση ήταν αυτά να προωθηθούν από τους ε, εκπροσώπους μας. Open Access Platforms για τις ε, μεταφορές σιδηροδρόμων και το ίδιο για τις δημόσιες μεταφορές και τους ε, τουριστικούς χώρους. Για την επιτροπολογία έχει κυκλοφορήσει το έγγραφο, για την οργάνωση της συναντήσεων των συντονιστών. Ναι, μεν να μπορούν να συμμετέχουν οι αναπληρωτές συντονιστές και οι αντιπρόεδροι, αλλά μόνο ένα συντονιστής αναπολιτική ομάδα να λάβει το λόγο και οι αντιπρόεδροι μόνο εφόσον τους καλέσει ο πρόεδρος. Και για τα διάφορα αυτά να καθίσταται γνωστά, να ανακοινώνονται μέχρι την πέμπτη το απόγευμα, ή μάλιστα το μεσημέρι, εκτός αν υπάρχει κάτι το κατεπήγον, οπότε ο πρόεδρος θα λάβει στην ουσία απόφαση εάν θα την θέσει υπόψη των συντονιστών. Στα διάφορα, οι συντονιστές έλαβαν υπόψη το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα. Έχει αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Χρειάστηκε να το κάνουμε διότι ε, έχει επιβάλει το Προεδρείο περικοπές στο κόστος της διερμηνίας. Για τις αντιπροσωπείες η αντιπροσωπεία για τις ΗΠΑ για το 2012 δεν προχώρησε το ταξίδι δηλαδή, της αντιπροσωπείας επίσης μας έχει προσκαλέσει, δηλαδή τους συντονιστές. Η ελβετική κυβέρνηση για τις 19 21 Σεπτεμβρίου για τις ακροάσεις. Σχέδιο προγράμματος για τις ακροάσεις για την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη 24 Απριλίου και για, επίσης για τις guidelines για τα δίκτυα στις 20 Μαΐου. Τώρα για Ηνωμένες Πολιτείες Ισλανδία, Νορβηγία. Οι συντονιστές είπαν να μην κάνουμε καμία δράση, να αναμένουμε την απόφαση του δικαστηριού, διότι έχει προσφύγει κατά του Συμβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η νομική επιτροπή του Κοινοβουλίου υποστηρίζει την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα αναμένουμε μέχρι ότου εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου πριν να αποφασίσουμε τι δράση θα αναλάβουμε για το διαρθωμένο διάλογο για το πρόγραμμα εργασιών 2013 της Κομισιόν οι πολιτικές ομάδες θα μπορούν να προτείνουν έναν περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων μέχρι τις 20 Απριλίου και θα συζητηθεί αυτή στην συνάντηση των συντονιστών του Απριλίου. Για το follow-up της έκθεσης Φιντάντσα για την ε, μόνιμη ομάδα εργασίας για τον τουρισμό αποφασίστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών να προεδρεύει της ομάδας εργασίας και να μπορεί να αναθέτει ε, δράσεις στον ίδιο τον κύριο Φιντάντζα. Οι αντιπροσωπείες, θα, οι πολιτικές ομάδες μάλλον, οι πολιτικές ομάδες θα ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέχρι τις 30 Μαρτίου και τα υπόλοιπα θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση. Αυτά λοιπόν για την συνάντηση των συντονιστών. Έχετε ερωτήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τα εγκρίνεται και προχωρώ στο επόμενο που είναι οι συζητήσεις για τη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κήτους για τα πετρελαιοφόρα. Κύριε Πρόεδρε, ο τριμερής διάλογος τελείωσε θετικά. Το Συμβούλιο θυγραμμίστηκε με τις θέσεις που ψηφίσαμε στην Επιτροπή. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε προς οριστική λύση σε πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια. Okay, thank you, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Ρίκε. Άρα έχει γίνει συμφωνία για πρώτη ανάγνωση στο τεχνικό επίπεδο για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κήτους για την Ολομέλεια αναμένεται να πάει τον Μάιο αυτή η συμφωνία πρώτης αναγνώσεως. Έχει καλώς λοιπόν και προχωρώ. Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση μελέτης για την μείωση της συγχωρήπανση των σιδηροδρόμων. Έχουμε λοιπόν κοντά μας σήμερα μια στιγμή να δώσω τις σημειώσεις. τους κυρίους Κλάους και Κοσιέκ, που είστε, και οι δύο του Fraunhofer Ινστιτούτου για εφοδιαστική και ροές υλικών. Θα θυμάστε ότι η European Environment Agency το 2010 μας είπε πόσα εκατομμύρια πολιτών επηρεάζονται από την ηχορύπανση κάθε μέρα, Και η Επιτροπή Μεταφορών αποφάσισε να αναθέσει πλήρη μελέτη για την ηχορύπανση των σιδηροδρόμων, κυρίως των σειρμών, των φορτηγών σειρμών, καθώς και αυτών που περιλαμβάνουν παλαιά ε, οχήματα ή και μηχανές Έλξεω. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στους κύριους Κλάους και 26. Ποιος πρώτος θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Κλάουσενς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, είμαι καθηγητή υπεύθυνο για τι μεταφορέ και επιμελητία στο Πανεπιστήμιο Ντότμοντ. Παρουσιάζω κοινή εργασία που κάναμε συναδέλφου στη Καλσλούη και στο Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ. Όσον αφορά την ηχορύπανση του σιδηροδρόμου, ξεκινούμε από την παρούσα κατάσταση. Ποιε είναι οι πηγέ τη ηχορύπανση του σιδηροδρόμου και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να μειωθούν τι οικονομικά κίνητρα μπορούν να δοθούν, τι ρυθμίσεις μπορούν να θεσπιστούν και πώς μπορούν να σχεδιαστούν οι καλύτερα δραστηριότητες όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος. Μια σημαντική ε, μειονότητα κατοίκων επηρεάζεται. 12 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη και έχουμε το όριο των 55 δεσιμπέλ ε, μέρα και νύχτα. Αυτό είναι ο περιβαλλοντικό θόρυβο. Και το βράδυ έχουμε χαμηλότερο επίπεδο, όριο, σαν όριο. Ξεκινάει στι 11 το βράδυ αυτή η περίοδο. Περίπου 9 εκατομμύρια κατοίκου ε, επηρεάζει ο θόρυβο. Τα κράτη-μέλη έπρεπε να δώσουν στοιχεία χαρτογράφηση θορύβων και διάφορα σχέδια δράση σχετικά. Σε πρώτερη ευρωπαϊκή νομοθεσία αυτό μα βοήθησε ε, να έχουμε μια καλή εικόνα όσον αφορά της εικόνας των θορύβων σε διάφορες κατοικήσιμες περιοχές και διάφορες περιοχές της Ευρώπης γενικότερα. Όσον αφορά τα μέτρα, κάποια μέτρα ξεπερνούν το τοπικό επίπεδο, θα αναφερθώ σε περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Τώρα βλέπουμε ποιος πληθυσμός επηρεάζεται. Δεν υπάρχει ίδιο ε, καταμερισμός ισότιμος όλη την Ευρώπη. 85% του πληθυσμού μένει στις μεγαλύτερες χώρες που έχουν και περισσότερη κυκλοφορία σιδηροδρόμων. Βλέπετε, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Και αν δείτε και τι γίνεται στις άλλες χώρες, η Σλοβακία, η Τσεχική Δημοκρατία και άλλες χώρες επίσης. Ε, εκεί υπάρχει σημαντικό, και εκεί υπάρχει ποσοστό πληθυσμού που επηρεάζεται. Βλέπουμε, λαμβάνεται υπόψη και η πυκνότητα του πληθυσμού, η δομή των δικτύων σιδηροδρομικών που έχουν κάποιες χώρες. Άρα, κάποιε χώρε τελικά έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλε όσον αφορά την ηχορύπανση. Βλέπετε εδώ στα ίδια στοιχεία, με άλλη χαρτογράφηση, βλέπετε το ποσοστό των πληθυσμών που πλήγεται σε κάθε χώρα. Η Αυστρία και η Σλοβακία είναι επικεφαλής λόγω τη σημασία που έχει σιδηροδρομικό τομέα στι χώρε αυτέ, τη γεωγραφία και τη όλη διάθρωση των συστημάτων. Οι πηγέ τώρα. Τρει πηγέ Μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα είναι ο ήχος του κινητήρα της μηχανής έλξης που δημιουργεί τον περισσότερο θόρυβο. Μετά από 30 200 χιλιόμετρα την ώρα είναι ο ήχος του σειρμού και επηρεάζεται βέβαια και από την επιφάνεια των τροχών, από την ποιότητα των τροχιών, των σιδηροτροχιών και σε πολύ μεγάλες ταχύτητες επίσης Έχουμε και τον αεροδυναμικό θόρυβο που έχει ένα ποσοστό όσον αφορά τους θορύβους. Ε, βλέπουμε άλλη μια εικόνα εδώ, παλαιότερους σειρμούς και ο σύγχρονους. Σύγχρονοι σειρμοί είναι αυτοί που κατασκευαστει 10-15 τελευταία χρόνια. Έχουμε μειώσει όσον αφορά τις μηχανές έλξης, ε, μείωση του θορύβου, αλλά η βιωσιμότητα των ε, όλων αυτών των αμαξοστοιχειών ε, η διάρκεια ζωής είναι μεγάλη. Μπορούμε να μειώσουμε το θόρυβο στην πηγή και στις υποδομές. Ε, θα επιστρέψω σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα φρένα. Ε, κάλυψη, ε, και προστασία των ε, μηχανών έλξεως, προστατεύουμε από το θορύβους, καλύπτουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, να αφορά τις Έχουμε δυνατότητες να βάλουμε διάφορους μηχανισμούς απόσβεσης κραδασμών, ε, να ψώσουμε τύχη για να μειώνεται η διάδοση θορύβου και θέμα συντήρησης των γραμμών επίσης. Είναι πολύ σημαντική συντήρηση για τη μείωση του θορύβου. μακρόν, είχαμε κάποια φρένα που χρησιμοποιούσαμε με τα κάκια που ε, δημιουργούσαν ε, με την τριβή ε, ανομαλίες στην επιφάνεια του, του, τροχού και αυτό κυρίως για τα φορτηγά τρένα δημιουργούσε αύξηση του θορύβου και μέχρι τώρα σχεδόν όλοι οι σειρμοί μεταφοράς εμπορευμάτων είχαν αυτά τα φρένα οπότε είχαμε υψηλότερα επίπεδα ηχορύπανσης από τα φορτηγά τρένα σε σχέση με τα επιβατηγά. Αυτά τα φρένα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τα επιβατικά τρένα και λιγότερο για τα εμπορικά τρένα γιατί κοστίζουν περισσότερο. Αντί για σίδηρο χρησιμοποιούμε άλλα υλικά τώρα στα φρένα και μειώσαμε κατά 8 περίπου το θόρυβο. Και το πώς είναι δομημένο το σύστημα των τροχών για τους μηχανισμούς απορρόφησης κραδασμών. Ε, τα μορτισέρ ε, βοηθούν, αλλά γίνεται πιο ακριβώς ο σύρμος τότε. Και νέοι μηχανισμοί για τους τροχούς υπάρχουν δισταγμοί να χρησιμοποιηθούν. Στο συνδρομικό τομέα, βλέπετε, ε, πρώτη στο ρόλο παίζει η ασφάλεια. Και η διάρκεια. Τα οικονομικά θέματα και ο θόρυβος είναι και αυτά σημαντικά στοιχεία. Από την Ιαπωνία βλέπουμε, εδώ αυτές τις φωτογραφίες, στην Ευρώπη έχουμε πολλούς σειρμούς υψηλής ταχύτητας που κινούνται μακριά από τις κατοικημένες περιοχές, είναι μικρότερο το πρόβλημα. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, προχωρώ και βλέπουμε αυτά τα φράγματα του στίχους για το θόρυβο μέχρι 2 μέτρα σε πολλές περιοχές σε ύψος και σε άλλα μέρη έχουμε μέχρι 5 μέτρα αυτούς τους στίχους και μπορεί να μειωθεί ο θόρυβος στο μήκος του σιδηροδρόμου, αλλά μειώνει τη θέα όμως. Συντήρηση των γραμμών, των σιδηροτροχιών, βελτιώνει πολύ το θόρυβο, άμα γίνει σωστή συντήρηση. Χρειάζεται ελίανση, τακτικά να γίνεται ελίανση για να μειωθεί ο θόρυβος που προέρχεται από τις ανομαλίες μεταξύ ε, τροχού και ράγας. Ε, αν βάλουμε σύνθετα υλικά στα φρένα, μειώνεται από τα τακάκια θόρυβος. Ε, διότι επηρεάζει λιγότερη ανομαλία που έχει η επιφάνεια του τροχού. Και έτσι μπορούμε σημαντικά να μειώσουμε το θόρυβο. Αλλά αφού τα περισσότερα βαγόνια αλλάξουν και βάλουμε το νέο υλικό και γίνουν πιο σύγχρονα. Αν βάλουμε το μισό εξοπλισμό με αυτά τα καινούργια ε, μηχανισμούς μόνο 30 δεσιμπέλ μειώνουμε το θόρυβο. Υπάρχει αισθητή διαφορά αλλά όχι μεγάλη. Ποιο είναι το βασικό όφελος. Με 90-95% αλλαγή του εξοπλισμού αν χρησιμοποιήσουμε νέα τεχνολογία ε, όσον αφορά ε, τους τροχούς και το σύστημα των τροχών. 95% τότε αλλαγή θα οδηγεί σε μείωση 12 δεσιμπέλ του θορύβου. Ε, είναι ένα πρόβλημα κυρίως με τις αμαξοστοιχίες μεταφοράς εμπορεύματος, όχι τόσο για τις επιβατικές ε, αμαξοστοιχίες. Διότι εκεί έχουμε καλύτερο κράμα σειρμών συγχρόνων και παλαιών. Όσον αφορά Έχουμε 370.000 μονάδες βαγόνια για μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα υλικά σε όλες. Κάναμε μελέτες και οι μελέτες δείχνουν ότι έχουμε 370.000 με 400.000 μονάδες στην Ευρώπη με τα κάκια τέτοια και αν αλλάξουμε το, τα συστήματα σε αυτά τα βαγόνια τότε μπορούμε με αποτελεσματικότατο τρόπο να μειώσουμε το θόρυβο, τον ηχορύπανση του σιδηροδρόμους διότι επηρεάζει κυρίως το βράδυ τον κόσμο ο θόρυβος. Και υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία, που... κόμβοι, όπου εκεί χρειάζονται ε, ιδιαίτερα μέτρα, συμπληρωματικά μέτρα. Όσον αφορά τα κίνητρα, πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να θεσπίσουν μέτρα για να οδηγήσουν σε μείωση του θορύβου και στις υποδομές και στην πηγή λαμβάνοντα μέτρα χωρί να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει μια γρήγορη λύση για την αποφυγή του θορύβου. Αν αποφα... φύγει κανεί τη μεταφορά μέσω σιδηροδρόμων, αλλά αυτό δεν ταιριάζει με τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ αποφάσει. Ε, και είναι και κάτι δυσάρεστο οικολογικά. Και θα έχει και οικονομικέ συνέπειε ε, σε αρκετού τομεί. Εμείς προτείνουμε εδώ κάποιο τέλος για πρόσβαση στις γραμμές με βάση το θόρυβο θα πρέπει να προβλέπετε να μπουν σύνθετα υλικά στα φρένα, θα πρέπει να, να δούμε επίπεδα χρηματοδότησης, να δώσουμε αρνητικά κίνητρα, θετικά κίνητρα και χρηματοδότηση. Τι γίνεται. Αυτά τα τέλη για το θόρυβο θα πρέπει να προβλέπουν μπόνους για σειρμούς που έχουν, δημιουργούν χαμηλό θόρυβο, λαμβάνοντα υπόψη τις δυνατότητε απώλειας ανταγωνιστικότητας των έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς, θα πρέπει να χρηματοδοτούμε και για ξεχωριστού σειρμού, ξεχωριστά βαγόνια, αλλά και ολόκληρου σειρμού να, να, χρηματοδοτήσουμε την αλλαγή του. Και θα πρέπει να καλύψουμε την αύξηση του λειτουργικού κόστου ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ανεξάρτητα από κάθε κράτο μέλο. άμεση χρηματοδότηση θα επιταχύνει την εισαγωγή νέων μηχανισμών με μειωμένο θόρυβο. Θα πρέπει τα μέτρα να βασίζονται να έχω σαν στόχο την πηγή του θορύβου. Αυτός ο θόρυβος, TSI, είναι κάποια όρια που καθορίζουν το θόρυβο που εκπέμπει ένας ερημός. Εάν αυτά τα όρια θα καλύπτουν και τους ε, φυστάμενους ηρμούς ή όχι, αν αυτά τα όρια που έχουμε θέσει καλύπτουν και τους παλιούς και τους πιο καινούριους φυρμούς. Πρέπει να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά τα θέματα, τι υποχρεώσεις υπάρχουν για εναρμόνιση τελών που θα καταβάλλονται για την παραγωγή θορύβου από τους σιδηροδρόμους, για να δημιουργηθεί αυτό το τέλος που θα εξαρτάται από το θόρυβο που παράγεται και θα πρέπει αυτοί που διαχειρίζονται τις υποδομές να συντηρούν τις υποδομές με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνουν το θόρυβο που θα παράγει ε, ε, ένα σύστημα το οποίο δεν συντηρείται σωστά. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα, ώστε τα κράτη-μέλη να πρέπει να εισαγάγουν τη σωστή χρηματοδότηση, να θεσπίσουν σωστή χρηματοδότηση για τοπικούς ιδεροδρόμους αλλά και διεθνείς ιδεροδρομικούς σιδηροδρομικούς σειρμούς. Για το θόρυβο TSI, σε κάποια... Σε 10-12 χρόνια θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά όχι σε 2-3 χρόνια για τεχνικούς λόγους. Σε 12 χρόνια θα λυθεί αν έχουμε υπόψη μας ότι οι συνέπειες για τον τομέα θα είναι ισορροπημένες, ε, ο ανταγωνισμός των σιδηροδρόμων έναντι των άλλων τρόπων μεταφορών παραμένει, δεν θα κινδυνεύσουν οι σιδηροδρόμοι και θα Πρέπει να γίνεται ένα ανταγωνισμό, ούτω ώστε να αμείβεται αυτό που έχει τι καλύτερε επιδόσει όσον αφορά τη μείωση του θορύβου από του φορεί. Ανταγωνισμό μεταξύ οδικών και συνδρομικών μεταφορών, κάτι πολύ σημαντικό. Αν επιβληθούν όρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω υπάρξει απομάκρυνση από του σιδηροδρόμου. Άρα πρέπει παράλληλα να κινηθούν τα μέτρα. Πέρα από τα οικολογικά μέτρα, που πρέπει να έχουν προτεραιότητα, θα υπάρχουν και κάποια σημεία δύσκολα τοπικά όπου χρειάζονται ειδικά μέτρα για τους σιδηροδρόμους που θα ταιριάζουν με τη σωστή χρηματοδότηση για τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών. Αυτά και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Okay. No, no problem. Uh, questions from κανένα πρόβλημα. Ποιος θέλει το λόγο για απορίες, Μάικλ και μετά οι υπόλοιποι. No, Mr. Kramer. Well, Mr. Kramer first and I... Πρώτα ο κύριος Κράμερ και μετά θα δω ποιοι άλλοι θέλουν το λόγο για να τους εγγράψω στον κατάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την διάλεξή σας. Εγώ είδα όμως να μου λείπουν κάποια νούμερα. Να ξέρουμε δηλαδή πόσο θα κοστίσει αυτή, αυτός ο εξοπλισμός. Εάν δηλαδή μπουν σε 80% των, βαγονιών, των φορτηγών βαγονιών στην Ευρώπη αυτά τα νέα φρένα θα είναι περίπου 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για 10 χρόνια θα είναι, ε, εκατομμύρια, συγγνώμη, θα είναι 350 εκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια είναι, προβλέπονται για την κατασκευή τείχων κατά των θορύβων. Το πρόβλημα στην ε, Ευρώπη είναι ότι δεν υπάρχει συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον του τροχαίου υλικού. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι, τα νούμερα που σας είπα είναι σωστά και θα συνιστούσατε όχι μόνο τις τιμές για την πρόσβαση στις, ε, ε <clears throat> στις, τροχές, στις ε, με κάποιο ειδικό τέλος, αλλά θα ήταν και καλύτερα. Αν μου επιτρέψετε θα σας απαντήσω και στα γερμανικά βεβαίως. Στην εκτενή μελέτη μας περιλάβαμε όλα τα νούμερα που ήταν διαθέσιμα. Οι τάξεις μεγέθους των βαγονιών είναι περίπου 380.000 και το κόστος επανεξοπλισμού είναι περίπου 2.000 ευρώ αναβαγώνει. Είναι βέβαια σημαντική πρόκληση αυτή, διότι καταλήγει κανείς σε 750 εκατομμύρια ευρώ περίπου για τον επανεξοπλισμό αυτό. Όπως λέτε όμως είναι λιγότερο δαπανηρό το μέτρο από ότι η κατασκευή ειδικών υποδομών ε, ε, για την μείωση του θορύβου. μια συμπλήρωση, κύριε Κράμερ, στη μελέτη μας, σε ένα σημείο της μελέτης μας, κάτι που δεν περιλήφθη λόγω της συντομίας της ε, προφορικής ε, διαλέξεως, έχουμε πανάκριβους τείχους για τη μείωση του θορύβου. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να λάβουμε άλλα μέτρα, ιδίως για την ε, κίνηση τη νύχτα. Είναι δυνατόν λοιπόν να ληφθούν κάποια χρήματα από την κατασκευή υποδομών και αυτό να γίνει και με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ, η κυρία Δερνιού. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγώ έχω ερωτήματα για το κόστος. Όπως είπατε, θα πρέπει να αναζητηθεί κοινοτική χρηματοδότηση για τα συνοδευτικά μέτρα και κυρίως ε, τις ε, μαύρες κυλίδες που θα μας στοιχήσουν πολύ ακριβά. Υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης από τα κράτη-μέλη. Ε, υπενήστε κάτι τέτοιο η μελέτη, αλλά από ό,τι ξέρω μόνο οι Γερμανία και κάτω χώρες έχουν δεσμευτεί για τέτοια χρηματοδότηση μέχρι στιγμής. Και μάλιστα για ποσά που δεν ξεπερνά το 50% των επενδύσεων. Επιπλέον η χρηματοδότηση θα πρέπει να καλύπτει φυσικά τις επενδύσεις, αλλά και το κόστος σχετικά με το κύκλο της ζωής των προϊόντων. Πιστεύετε ότι μπορούν να βρεθούν κάποιες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα κράτη-μέλη προσπαθούν για προφανείς οικονομικούς λόγους να περικόπτουν να περικόπτουν συνέχεια τις δαπάνες τους. Ευχαριστώ. Όπως ε, είπατε σωστά, ελάχιστες είναι οι πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει από τα κράτη-μέλη. Ακόμη και στη Γερμανία υπάρχει τέτοια πρόθεση θεωρητικά, αλλά ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί σε ένα νομοθετικό κείμενο. Φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνουν τα κράτη-μέλη πόσος κόσμος επηρεάζεται από κάτι τέτοιο. Και μπορεί το πρόβλημα να λυθεί σε 25 χρόνια, αλλά αν θέλουμε να το λύσουμε νωρίτερα, σε μία δεκαετία, θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερα κονδύλια στις επενδύσεις, γιατί ο ίδιος ο κλάδος δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Δεν υπάρχουν πελάτες που θα συμφωνήσουν να πληρώσουν ένα συμπλήρωμα στο εισιτήριό τους επειδή χρησιμοποιείται κάποιος εξοπλισμός για την μείωση, των περιορισμών του θορύβου. Είπαμε ότι θα ήταν πρόκληση να βρεθούν νομοθετικές προτάσεις για συγχρηματοδότηση κοινοτική και εθνική. Εμείς μπορούμε απλώς να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να προτείνουμε κάποιες λύσεις, αλλά δεν μπορούμε να τις δώσουμε εμείς τις λύσεις. Ο κύριος Γκάλερ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης και εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα. Συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ ότι θα ήθελα και εγώ περισσότερα νούμερα. Είπατε όμως ότι ε, περιλαμβάνεται στην πλήρη έκδοση της μελέτης σας. Νομίζω πολιτικά αντιμετωπίζουμε την αναγκαιότητα της ανάληψης δράσης για να γίνει περισσότερο αποδεκτή και όλα η μεταφορά των εμπορευμάτων από τον κόσμο. Στην δική μου εκλογική περιφέρεια περνάει αυτός ο μεγάλος διάδρομος από Τζένοβα στο Ρότερνταμ και μάλιστα και αριστερά και δεξιά είναι βουνά και δεν υπάρχει απαγόρευση κίνησης των τρένων τη νύχτα αντίθετα από τα αεροπλάνα και εκεί πραγματικά έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ ο κόσμος αν ακούσουν και τα νούμερα πώς θα αυξηθεί δηλαδή η κίνηση των ε, σύρμων δεν θα υπάρξει αποδοχή αν δεν κάνουμε κάτι και μάλιστα ως το δυνατόν ταχύτερα και ως το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Η ερώτησή μου προκειμένου είναι η εξή, γιατί εσείς εξηγήσατε τα διάφορα μέτρα, τι μπορεί να κάνει κανείς δηλαδή. Πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατό εάν υπάρξει διευρωπαϊκά μια προσπάθεια ώστε για την έγκριση κυκλοφορίας νέων βαγονιών, τα νέα φρένα που είπατε κτλ. Δηλαδή αν πούμε ότι δεν έχουμε λεφτά για να τροποποιήσουμε τα συστήματα πέδησης όλων των βαγονιών, όταν όμως γίνεται αγορά νέων βαγονιών, τότε η διαφορά στην τιμή μεταξύ της παλαιάς, ε, του παλαιού τρόπου πέδησης και του νέου ίσως δεν είναι τόσο σημαντική. Μήπως λοιπόν αυτός είναι ένας τρόπος να επιβάλλουμε δηλαδή την προδιαγραφή αυτή για την αγορά νέων βαγονιών και μετά για να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού πανευρωπαϊκά να πούμε ότι θα προβλέψουμε χρονικά μία φθήνουσα στήριξη, δηλαδή όποιος κάνει τις τροποποίησεις αυτές τα βαγόνια νωρίτερα θα, θα λαμβάνει περισσότερη στήριξη και όποιος αργότερα, λιγότερα και ούτω καθεξής βρίσκεται ότι αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί, να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν έχω επαρκή εμπειρία για να κρίνω εάν όντω μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά νομίζω ότι θα αποφευγόταν με τον τρόπο αυτό κάποια στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσα στην Ευρώπη. Ο εμπειρογνώμων ευχαριστώ, κύριε Γκάλερ, για την ερώτηση. Εσείς είπατε με απλούστερα λόγια αυτό προσπαθήσαμε να πούμε εμείς στη μελέτη, διότι υπάρχουν επιμέρους πτυχές που έχουμε γράψει κιόλας ότι εγκρίνονται τώρα η κυκλοφορία μόνο των νέων βαγονιών και η TSI που αναφέρεται στον θόρυβο των ε, βαγονιών, τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας δηλαδή, εάν αυτό τώρα μπορεί να διευρυνθεί για να περιληφθούν και τα νέα συστήματα πέδησης, τότε βέβαια θα είναι λιγότερο θορυβόδη τα τρένα αυτά. Αλλά ίσως προς τα εκεί πρέπει να κατευθυνθεί. Όπως και στις οδικές μεταφορές με την μείωση εκπομπών ρήπων των κινητήρων, είπαμε ότι μπορεί να, μπορεί να επιβληθεί ένα όριο που πρέπει να τηρηθεί και από εκεί και πέρα να υπάρχει μια επιβάρυνση. Το σημαντικό είναι όταν μιλεί κανείς για κόστος πρέπει να φροντίσουμε ώστε να μην υποστεί βλάβη η ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων με την υπερβολική επιβάρυνση με τέλη και διάφορα άλλα. Το, είναι προτιμότερο δηλαδή να βασιστεί σε ένα σύστημα μπόνους και όχι σύστημα μπόνους μάλους. Βέβαια και η τεχνολογία μπορεί στο μεταξύ να αλλάξει. Η κυρία Μάισνερ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Μιχαήλ Γκάλερ. Και βέβαια συζητούμε τώρα για παράδειγμα για τον θόρυβο των αεροσκαφών και απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων και ξέρουμε τι σημαίνει η προσπάθεια μείωσης του θορύβου από τις μεταφορές. Ο θόρυβος μπορεί να οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Και βέβαια η κυκλοφορία όλων των μέσων μεταφοράς αυξάνεται. Νομίζω σωστά τα παρουσιάσατε τη μελέτη σας και η πρόταση του κυρίου Γκάλερ μου φαίνεται σωστή, δηλαδή να θεσπιστούν κάποια κίνητρα. Ίσως είναι μια καλή παραλλαγή αυτή, δηλαδή μια επιβράβευση, επιβράβευση αυτών που προβαίνουν σε επενδύσεις. Η ερώτηση για τα νούμερα σας ετέθη ήδη. Μας τα είπατε εμάς, είπατε και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως κοινοβούλιο για να παρακινήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση. Παρουσιάστε τη μελέτη σας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι συνήθως εδώ η διαδικασία έχει ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στη βάση των εμπειριών που συλλέγει και αυτή είναι άλλωστε αρμοδία να φροντίσει να μειωθούν οι ε, βλαβερές επιπτώσεις των περιβάλλων. Θα απαντήσω στα αγγλικά. Καταρχήν, ανταποκριθήκαμε σε ένα αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δώσαμε πληροφορίες που αντλήσαμε από επιστημονικές πηγές και από συνάντηση με εμπειρογνώμονες. Το επόμενο βήμα θα ήταν να μιλήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να παράσχουμε και σε αυτήν σύμβουλες. Έχω και εγώ μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Φιλομέτρησα την μελέτη και βρήθη πληροφοριών ε, για τη Γερμανία, την Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πού είναι οι πληροφορίες για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την ε, Ανατολική Ευρώπη, τις χώρες της Βαλτικής. Υπήρξε πρόβλημα με την ε, συγκέντρωση στοιχείων από τους σιδηροδρόμους αυτών των χωρών για το τι είδου ε, τροχαίο υλικό χρησιμοποιούν, τι είδου ε, συστήματα πέδησης χρησιμοποιούν. Γιατί όταν βλέπουμε 3.000 νέα σύγχρονα φρένα και 3.000 πεπαλαιωμένα, δεν νομίζω ότι είναι η ισότιμη κατανομή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι ξέρω, στον Ηνωμένο Βασίλειο τα περισσότερα βαγόνια, τα περισσότερες ε, αμαξοστοιχίε έχουν σύγχρονα συστήματα πέδησης. Αλλά πού βρίσκονται τα πιο απερχιωμένα συστήματα. Φαντάζομαι κάποιοι σιδηρόδρομοι τη Ευρώπης έχουν αυτά τα παλιότερα ε, συστήματα πέδησης. Ήταν δύσκολο να συγκεντρώσετε πληροφορίε για τις χώρες Ανατολική Ανατολικής Και αν ναι, τι στοιχεία έχετε για το ύψο του θορύβου στις χώρες αυτές. Όπως διαπιστώσατε, υπάρχει διαφορετική ποσότητα πληροφοριών ανάλογα με τις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Διαφέρει και η πυκνότητα των ε, σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων από χώρα σε χώρα. Άλλωστε, η μελέτη ξεκίνησε από χώρε που ενδιαφέρονται περισσότερο για το θέμα αυτό. Υπήρχαν περισσότερε δημοσιεύσει, υπήρξε μεγαλύτερη ανησυχία. Αν δείτε όμω τι σελίδε 33 έω 39 τη μελέτη, διαπιστώνεται ότι περιλαμβάνονται στοιχεία για τις δράσεις που αναλύθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν σιδηροδρόμους φυσικά και διαπιστώνεται ότι έχουμε στοιχεία και για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπάρχει ένα ποσοστό των πληροφοριών που αφορά αυτές τις χώρες. Για την Τσεχική Δημοκρατία, για παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι οι νέες σιδηροδρομικές γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τείχους θορύβου για τα 150 χιλιόμετρα. Επίσης στην Βουλγαρία υπάρχουν επίσης στοιχεία για τέτοιου ε, τείχου ε, περιορισμού του θορύβου, αλλά δεν υπάρχουν πολύ ακριβή στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την ένταση του σιδηροδρομικών μεταφορών, τον αριθμό των ε, προσώπων που επηρεάζονται, το υλικό που έχει δημοσιευθεί, υπάρχει όντως ανισορροπία. Για ορισμένες χώρες έχουμε πολλά στοιχεία και για άλλες πολύ λίγα. Κύριο Κράμερ. Ήθελα να μάθω και το εξή. Η Ελβετία παίρνει ανα, ε, πώς να πω, καθαρίζει τις γραμμές, τις λιένει τις ε, σιδηρογραμμές κάθε δύο χρόνια και όχι κάθε έξι χρόνια. Τώρα, επίσης, η νέα αυτή η πέδηση όμως ε, οδηγεί σε μεγαλύτερες φθορές των τροχών. Αυτό τι επίπτωση μπορεί να έχει. Τώρα, τα νέα βαγόνια, οι ε, αγορές νέων βαγονιών είναι περίπου 1 με 2% τον χρόνο. Αλλά αυτό που προτείνατε, ένα συνδυασμό δηλαδή, η Ελβετία είπε από το 2020 τα βαγόνια που κάνουν θόρυβο απαγορεύονται. Να πούμε και εμείς το ίδιο. Αυτός που θα αρχίσει πρώτος να αντικαθιστά θα πάρει και τις περισσότερες επιχορηγήσεις. Αυτά βέβαια θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα επιβάλλουμε στους ε, της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Βέβαια, εμεί δεν είμαστε η μοναδική εξουσία εδώ στην Ευρώπη, είμαστε μία από τι τρει. σω πρέπει να πάτε να τα πείτε και στου άλλου δύο. Να ξεκινήσω με το τελευταίο σχόλιο. Αν επιβάλλεται νομοθεσία που απαγορεύει τις ε, παλιές, ε, τους παλιούς σύρμους ε, μεταφοράς εμπορευμάτων και χωρίς άλλα κίνητρα και χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση, δεν θα έχουμε εξυγχρονισμό ε, των ε, σειρμών. Αντίθετα θα έχουμε μία μεταβίβαση των εμπορικών μεταφορών από τους σιδηροδρόμους στις οδικές μεταφορές, αν δεν υπάρχουν συμπληρωματικά κονδύλια και ενάψματα. Και πιστεύω ότι στις κατευθυντήριε γραμμές θα πρέπει να συμπεριλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και χρηματοδότηση και κονδύλια για να ε, γίνουν επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα περιορισμού του θορύβου. Σε ό,τι αφορά το τεχνικό σκέλος, Ισχύει αυτό που λέτε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είναι πλήρως λειτουργικό. Συνεχίζονται οι δοκιμές και μάλλον θα χρειαστεί κάποιος χρόνος ακόμη. Το κόστος αυξάνεται. Δεν μπορώ να σας δώσω όμως συγκεκριμένο αριθμό για το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος. Η Σουηδία ε, έχει, είναι πρωτοπόρα και στη χρηματοδότηση και στη συντήρηση. Αλλά δεν, ε, δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες οικονομικές πολλές χώρες μέλη να κάνουν αυτό που κάνει η Σουηδία. Μία άλλη ερώτηση. Η ε, αλληλεπίδραση σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Στη μελέτη σας σε ό,τι αφορά την κατάσταση των σιδηρογραμμών και την κατάσταση των τροχών ε, για το θόρυβο, ποια επιρροή τους ε, ή αντίστοιχα τα επίπεδα λάστιχα στο δρόμο. Έχετε στοιχεία για το πώς επηρεάζει η κατάσταση αυτών των στοιχείων το ύψος του θορύβου. Έχουμε εξετάσει διάφορες πτυχές στη μελέτη. Για παράδειγμα, μιλήσαμε για την αντικατάσταση των συστημάτων παίδησης από τα σιδερένια σε σύνθετα, όπως άλλο σύνθετο υλικό, όχι από σφύριλα το σίδερο. Αυτό το λάβαμε υπόψη στη μελέτη και αυτό που είπε ο κύριος Κράμερ, οι ε, εταιρείε που συντηρούν τι υποδομέ είναι υποχρεωμένες να συντηρήσουν και τι γραμμέ. και ε, φαντάζομαι υπάρχουν διάφορα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό σε τοπικό επίπεδο. Πάντως ε, λάβαμε υπόψη και τις διατυχές του ζητήματο. Άλλο... Άλλος κανείς, άλλα σχόλια υπάρχουν. Όχι, ευχαριστώ τους δύο εμπειρογνώμονες για την παρουσίαση της μελέτης και για την απάντηση που δώσατε στις απορίες των συναδέλφων. Φαντάζομαι τα μέλη της Επιτροπής θα διαβάσουν με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη μελέτη σας. Σας ευχαριστώ. Next item on the agenda is Επόμενο σημείο της σας διάταξης, τα διάφορα. Δεν υπάρχουν όμως. Προσοχή συνεδρίαση. Στις Βρυξέλλες, ημέρα Δευτέρα, 23 Απριλίου, στις 3 το απόγευμα. Λύεται η συνεδρίαση, αλλά παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν για τη συνεδρίαση του μαύρου, της μαύρης λίστας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τους υπόλοιπους ε, η συνεδρίαση τελειώνει.